Ε, με τα πρώτα με τις, ε, ε, πρώτες, τα πρώτα σημεία της ημερήσης Η κυρία Παλιαδέλη είπε ότι δεν θα είναι με παρούσα αύριο για προσωπικά ζητήματα, ούτε και σήμερα η κυρία Μπρούνη για θεσμικούς λόγους. Σας ενημερώνω ότι όσον αφορά την αναφορά στο σημείο 7 θα είναι παρόν ο παραγωγός γιατί μιλάμε για ένα θέμα που αφορά την εμπορευματοποίηση μιας κρέμας και έχει ζητήσει να είναι παρόν ο αναφέρον. Τα, επίσης θα είναι παρόντες οι αναφέροντες για τα σημεία 11, 12, 13 και 14. Ε, αύριο το πρωί για την έκθεση της αποστολής ΒΕΛΒΑ θα είναι παρούσες οι Ισπανικές Αρχές της επαρχίας ε, ΒΕΛΒΑ καθώς και οι αναφέροντες υπό ε, κατόπιν ετήματος της κυρίας Γρούνη. Ωστόσο θα το συζητήσουμε γύρω στις 11 γιατί η κυρία Γκρούνη ταυτόχρονα έχει ε, ένα θέμα στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ζήτησε να καθυστερήσει λίγο η εξέταση αυτού του σημείου. Αύριο από τις 11 θα έχουμε ψηφοφορία για την έκθεση του συναδέλφου Τουργκάης για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών και ε, στη συνέχεια θα ψηφίσουμε την ε, γνωμοδότηση για τη βιοπικιλότητα της συναδέλφου Μποστινάρο. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη θα θεωρήσουμε πως εγκρίνεται. Στη συνέχεια θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης 26 και 27 Απριλίου. Ούτε γι' αυτό υπάρχουν αντιρρήσεις, οπότε θεωρούμε πως εγκρίνονται. Ε, Ήθελα να σας ενημερώσω ότι η διαδικασία συνεργασίας, ενισχυμένης συνεργασίας με βάση το άρθρο 50 του κανονισμού σε σχέση με την έκθεση για την λαϊκή πρωτοβουλία έχει περάσει κάποιες στιγμές αβεβαιότητας στη φάση εξέτασης από, την, από πλευράς της Προεδρίας, όμως τελικά καταφέραμε να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα, γιατί υπήρχαν δηλαδή κάποιες αντιρρήσεις τεχνικής φύσης για τη διαδικασία που ακολουθήσαμε. Τώρα έχουμε ως ε, μόνη προσαρμογή που θα πρέπει να γίνει, γιατί επιτύχαμε την έγκριση από πλευράς του Προεδρίου θα πρέπει λοιπόν να επικυρώσουμε την απόφαση ένδειξης, υπόδειξης μάλλον του εισηγητή, απόφαση που έχουμε λάβει σε μια προηγούμενη φάση, πριν δηλαδή να έχουμε την άδεια. Μόνο για διαδικαστικούς λόγους λοιπόν θα πρέπει να επικυρώσουμε τον εισηγητή και αύριο θα το κάνουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Όπως για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ε, αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις όσον αφορά τις αναφορές που συμπεριλαμβάνονται σε εκείνο το προσάρτημα, θα έχουν θα θεωρηθεί ότι κλείνουν αυτές οι αναφορές. Εάν υπάρξουν αντιρρήσεις θα, θα περάσουν στο σημείο α της ημερήσιας διάταξης. Τώρα, η πρώτη αναφορά που έχουμε να εξετάσουμε είναι η 5, ε, το σημείο 5, 986 κάθετος 2006 που έχει υποβάλει ο Θεόδωρος Δαλμάρης, δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Οπότε θα δώσω άμεσα το λόγο στον υπεύθυνο της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην Μαγκαλή Λενοέλ. Oui. Bonjour, euh, madame et monsieur les députés. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις, για αυτήν ε, την ε, αναφορά που θα σας θυμίσω ότι αποτελεί και ε, αντικείμενο καταγγελίας. Η διαδικασία έρευνας που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά τις επτά ε, ε, εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν χωρίς έγκριση και χωρίς σεβασμό στους κανόνες του υγειονομικούς στο παλιό τμήμα της ε, κρεαταγοράς του Ρέντι. Οι ελληνικές αρχές θεωρείται πως δεν τήρησαν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες και ζητήσαμε από τις ελληνικές αρχές να μας δώσουν τις παρατηρήσεις τους προς αυτό, ως προς αυτό το θέμα η Επιτροπή έλαβε μια απάντηση από τις ελληνικές αρχές 30 Απριλίου 2010. Σε αυτήν την απάντηση οι ελληνικές αρχές ενημέρωναν για την απόφαση των ε, κτηνιατρικών υπηρεσιών να αναστήλουν από τις 3 Μαρτίου 2010 την λειτουργία 7 καταστημάτων που εξακολουθούσαν να λειτουργούν στο παλαιό τμήμα της αγοράς του Ρέντι. Τελευταία έγινε μια αποστολή της ΟΑΒΕΣ τον Μάιο του 2010 και στο πλαίσιο αυτής της ε, αποστολής οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Κομισιόν πως κανένα κατάστημα δεν λειτουργεί πλέον στην παλιό τμήμα της αγοράς του Ρέντι και διευκρίνησαν ότι δύο από αυτά τα καταστήματα έκλεισαν και πέντε άλλα μεταφέρονται, είναι στη διαδικασία μεταφοράς στο νέο κομμάτι της αγοράς. Η Επιτροπή έχει την πρόθεση να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να επιβεβαιώσουν αυτές τις ε, πληροφορίες. Επιπλέον αυτή η αναφορά ε, αναφερόταν στην κατάσταση άλλων κρεταγορών στην Ελλάδα όπως αυτή του Ρέντι αλλά και το σφαγείο της Πρέβεζας. Ως προς αυτό, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν ε, την Κομισιόν από πλευρά του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων ότι αυτό το σφαγείο έχει πλέον κλείσει. Αυτά ισχύουν λοιπόν για το σφαγείο της Πρέβεζας ε, ε, θεωρείται ότι έχει κλείσει και όσον αφορά τα επτά καταστήματα που ήταν το αντικείμενο της έρευνας της Επιτροπής δεν λειτουργούν πλέον στην ε, παλαιά, στα παλαιά κτίρια της αγοράς του Ρέντι αλλά η Κομισιόν θα ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να επιβεβαιώσουν αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, άκουσα με πολύ προσοχή την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ε, είχα και εγώ έτσι ε, ε, έκανα τις έρευνές μου και ζήτησα πληροφορίες και όντως με πληροφορούν και μένα ότι από τις 7 επιχειρήσεις που είχαν μείνει ε, στην κρεαταγορά του Ρέντι, από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία που μου έχουν δώσει εδώ συνεργάτες μου, ε, πέντε έχουν μετεγκατασταθεί και δύο έχουν κλείσει οριστικά. Επίσης, με πληροφορούν ότι στις 19 Μαΐου του 2010, έχει σημασία που το λέω την ημερομηνία, ίσως μας βοηθήσει, στις 19 Μαΐου του 2010, κατά την καταληκτική συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του Γραφείου Τροφίμων και Εκτινιατρικών Θεμάτων και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμοδίων ελληνικών αρχών, ε, γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή αυτή η εξέλιξη. Και όσον αφορά το σφαγείο πρέβεζας, από τα στοιχεία που έχω μαζέψει, βλέπω ότι ε, έχει τελειώσει η υπόθεση της πρέβεζας και μάλιστα ε, έχω την πληροφορία ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας πήρε απόφαση το χώρο που λειτουργούσαν τα σφαγεία να τον κάνουν δημοτικό πάρκο. Ε, δεν ξέρω, προβληματίζομαι ε, μήπως θα έπρεπε να τελειώσει το θέμα αυτής της, ε, ε, πώς να το πω, της ε, έκθεσης, της αναφοράς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ε, τις ίδιες πληροφορίες που σας έδωσε η κυρία Ράπτη, τις έχω και εγώ και επιπλέον έχω την πληροφορία ότι υπάρχει και δικαστική απόφαση υπαριθμόν 9151 του 2009 απόφαση του 29ου τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίπτεται η αγωγή που είχε κάνει ο αναφέρον κύριος Δαλμάρης για την ίδια υπόθεση. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, οι ελληνικές αρχές πήραν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτιάσεων και στην περίπτωση της παλαιάς κρεβαταγοράς του Ρέντι και του σφαγίου της Πρέβεζας και ίσως θα πρέπει να μην δοθεί συνέχεια και να τεθεί πλέον ε, στο αρχείο η αναφορά του αναφέροντος. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ζητείτε να κλείσουμε το θέμα. Αν και η εκπρόσωπος της Κομισιόν μας είπε πως περιμένει ακόμα την οριστική έκθεση από πλευρά των ελληνικών αρχών. Άρα... Λάβαμε ένα σημείωμα αλλά που ακόμα είναι στην μετάφραση, αν κατάλαβα καλά. Εν πάση περιπτώσει, ίσω ε, για λόγου ορθότητα, ε, καλύτερα είναι να το κλείσουμε στο τέλο όταν θα έχουμε λάβει αυτή την επίσημη απάντηση και θα έχουμε και τη μετάφραση του σημειώματο που μα έφτασε ε, για να γνωρίζουμε ακριβώ με ποιο τρόπο θα κλείσει η αναφορά. Γιατί υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να επαληθευτούν, κύριε Ράπτη. Ε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο πάλι. Ε, με αφορμή την σημερινή συζήτηση, ε, θέλω να πω ότι βρεθήκαμε προ μιας ευχάριστης εκπλήξεως. Είδαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας να είναι όχι μόνο σε ίσο πώς να το πω, σε ίσο επίπεδο πληροφόρησης, αλλά να είναι ίσως και ένα κλικ πιο μπροστά ε, βεβαίως έχετε πάρα πολύ δίκιο, πρέπει να γίνουν όλα τυπικά, να είμαστε εντάξει και να περιμένουμε ε, και την επιβεβαίωση της Επιτροπής και να εκφράσω μια ευχή. Αυτή την ευαισθησία που επέδειξε σήμερα η Επιτροπή ε, δια της εκπροσώπου να την επιδεικνύει πάντα και σε όλα τα θέματα. Θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τους πολίτες της Ευρώπης. Αυτή την έκκληση προς την Κομισιόν την κάνουμε πάντοτε και καλό είναι να το επαναλάβουμε και με αυτή την ευκαιρία. Να διευκρινίσω για την ε, το θέμα των σχέσεων μεταξύ Επιτροπή και Κοινοβουλίου ότι η υπηρεσία μου μας ενημέρωσε για το ότι ε, λάβαμε άμεσα την απάντηση και εμείς, απλώς δεν έχει μεταφραστεί. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι είμαστε ισότιμοι ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να περιμένουμε μόνο να μεταφραστεί. Έφτασε στα ελληνικά, οπότε όπως φαντάζεστε δεν μπορώ εγώ να τη διαβάσω όπως φαντάζεστε χωρίς μετάφραση. Εγώ οφείλω να ανακοινώσω αυτή την απάντηση που λάβαμε και στους υπόλοιπους βουλευτές της Επιτροπής και μετά να κλείσει. Ο Ντέιβιντ μου ενημερώνει ότι πρέπει να περάσουμε στο σημείο 7, γιατί ο υπεύθυνο για την προηγούμενη, την 6, δεν είναι παρόν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη. Οπότε α πάμε στην 7. Είναι τρει αναφορέ μαζί. Τι έχουν υποβάλει η Μπίργκιτ Μέγερ, η Σίλβια Ρόγγελε και ο Ιβάλτραουτ Κούρτ γερμανικής ηθαγένειας. Ε, εδώ είναι παρόν ο παραγωγός και έχει ζητήσει το λόγο, όχι αναφέρωσες. Θα δώσω το λόγο στον ε, παραγωγό, στην παραγωγό, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Είμαστε από, μεταξύ αρκετών παραγωγών για, που ασχολούνται με την παραγωγή τέτοιων ε, προϊόντων, κρεμών και άλλων καλλιτικών προϊόντων ε, με, με φίλτρα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία. Προσπαθούμε λοιπόν να διατηρήσουμε, να εξασφαλίσουμε την ε, προστασία των ε, πολιτών και μέχρι στιγμής οι κρέμες αυτές δεν, έχουν, δεν περιλαμβάνουν διοξείδιο του τιτανίου. Προσπαθούμε λοιπόν ε, να δούμε τι γίνεται με όσους, ε, προσπαθούν, όσους θέλουν ακόμη να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ε, κρέμες γιατί αυτές έχουν αποδειχθεί ότι είναι βλαβερές για την υγεία και δεν υπάρχουν Ε, Έχουμε, λοιπόν, θέλουμε μια, μια εξαίρεση για τέτοια προϊόντα που έχουν βάσει την φυσική προστασία από τον ήλιο. Καταρχήν είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μιλούμε για σύσταση της Κομισιόν εδώ η οποία όμως είναι δεσμευτική. Το ΔΕΚ το επιβεβαιώνει αυτό και εκτός αυτού δείχνει η πράξη ότι τον η πρακτική στις καθημερινή, στην καθημερινή δουλειά των ευρωπαϊκών αρχών ότι όντως είναι πολύ, ότι δείχνει αρκετά μεγάλη δέσμευση όλο αυτό. Και επίσης το νέο πρότυπο που αναφέρεται έχει ε, λαθασμένη σχέση μεταξύ των ε, ε, ακτινών ε, UVA και UVB. Και τα φίλτρα αυτά δεν περιλαμβάνουν τις απαραίτητες, τα απαραίτητα στοιχεία για την προστασία. Και γι' αυτό, επειδή ο στόχος μας είναι πάντα η ύψιστη προστασία του καταναλωτή, και αυτό θα πρέπει να είναι και ο στόχος των, του κλάδου των, των καλλιτικών, ε, να θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτό προς το παρόν θεωρούμε ότι δεν εξασφαλίζεται η ε, προστασία δηλαδή, γιατί υπάρχουν και ε, κρέμες οι οποίες αφορούν παιδιά, που τις χρησιμοποιούν μικρά παιδιά και που δεν περιλαμβάνουν όλα αυτά τα φίλτρα φυσικής προστασίας. Μιλούμε δηλαδή για 10% που αποσύρθηκαν από την αγορά τέτοιων προϊόντων. Οπότε η παραγωγή θεωρούμε ότι δεν είναι ανάλογη και θα πρέπει να υπάρξει εξαίρεση. Τους λόγους τους είπα και να, να τελειώσω λέγοντας ότι ε, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ σήμερα. Είναι ένα βήμα προς τα μπρος για την ε, βιομηχανία καλλιτικών, αλλά Φυσικά είναι σημαντικό να μην περιοριστούμε μόνο στις ε, ε, αποσύρσεις από την αγορά προϊόντων, αλλά να έχουμε ως στόχο την, ε, τον καταναλωτή πάντα. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό. Και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Ο, η εκπρόσωπος, ο της Ρόμαν Μόκρη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Ήρθα εδώ για να σας εξηγήσω μερικά πράγματα όσον αφορά αυτές τις αντιλιακές κρέμες. Έχοντας ακούσει τις διαμαρτυρίες ε, της παραγωγού όσον αφορά την σύστασή μας, θέλω να υπογραμμίσω ότι η οδηγία αυτή δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στα φυσικά και τα χημικά συστατικά. Συνεπώς δεν υπάρχει νομική βάση εδώ για να πούμε ότι ένα, μια αντιλιακή κρέμα είναι με φυσικά συστατικά και μια άλλη με χημικά τέτοια. Δεν κάνουμε αυτή τη διάκριση. Φυσικά υπάρχουν διάφορες ιδιωτικέ πρωτοβουλίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τεθούν κριτήρια για να γίνεται η ταξινόμηση των ε, κρεμών είτε σε φυσικές είτε σε εκείνες που περιέχουν χημικά συστατικά. Τέτοια κριτήρια όμως, τέτοια σήμανση δεν αποτελούν μέρος της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τα καλλιντικά. Δεύτερον, η αποτελεσματικότητα των αντιλιακών κρεμών είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 ενέκρινε τη σύσταση για την αποτελεσματικότητα των αντιλιακών προϊόντων και των ε, κρεμών εκείνων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ελάχιστα συστατικά ουσιών που επιτρέπουν την προστασία από την ακτινοβολία α και β. Οι συστάσεις 1 3 για την ακτινοβολία αυτή διασφαλίζει ότι τα αντιλιακά προστατεύουν αποτελεσματικά από την ακτινοβολία αυτή. Υπάρχει μια αναλογία η οποία ε, δικαιολογείται, εξηγείται επιστημονικά από τα ποσοστά κτηνοβολίας που παίρνει το δέρμα και έχουν γίνει πειράματα εν vivo. Τρίτον, από πλευράς νομικής, όπως ήδη ακούσαμε, η σύσταση δεν είναι δεσμευτική νομικά. Και γι' αυτό είναι περίπλοκο να πούμε ότι κάνουμε εξαίρεση από τι τελικά, από μια σύσταση. Άρα εξαρτάται από τον ίδιο τον παραγωγό να αποφασίσει κατά πόσο θα συνεχίσει να παράγει ένα προϊόν φυσικό ή όχι. Θέλω επίσης να σας πω ότι μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία πληροφορία για το ότι η εφαρμογή της σύστασης έχει οδηγήσει καταναλωτές ε, με αλλεργίες σε υψηλότερα επίπεδα κινδύνου. Αυτή είναι η δικιά μου απόψη. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει συζήτηση και να δούμε κατά πόσο η παραγωγός μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και τις δύο απόψεις και τις σκέψεις της Κομισιόν για την ασφάλεια των καταναλωτών και από την άλλη τις ανησυχίες, τις σκέψεις των παραγωγών οι οποίες επίσης βασίζονται σε ένα πολύ ε, ευαίσθητο θέμα και ε, αφορούν μια μεγάλη ομάδα καταναλωτών. Έχουμε 80 εκατομμύρια αλλεργικούς στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι συσχετισμοί μεταξύ αυτών των καταναλωτών και των αλλεργιών που υπάρχουν. Το δέρμα είναι το πιο ευαίσθητο όργανο του ανθρώπου. Όλες οι χημικές ουσίες που α, περνάνε από το δέρμα καταλήγουν στο σώμα μας. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το α, ξεκαθαρίσουμε. Ας πούμε ένα παιδάκι μικρό που είναι στο νηπιαγωγείο εγώ ξέρω πολλά τέτοια παιδιά που ε, δεν τους επιτρέπεται στα... Οι γονείς δεν επιτρέπουν στα νηπιαγωγεία να τους βάζουν οποιοδήποτε προϊόν που να έχει χημικά προϊόντα, ε, χημικές ουσίες μέσα. Για να μπορέσουμε να ε, ε, αυξήσουμε την ασφάλεια και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την πρόσβαση σε φυσικά καλλιντικά. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα σχετικά με αυτό που είπε μόλις η συνάδελφος. Το δικό μου πρόβλημα είναι το εξή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε επισήμανση για να λύσουμε το πρόβλημα. Αν κατάλαβα καλά, η κρέμα δεν είναι βλαβερή. Έχει προστασία από τον ήλιο, από τις ηλιακές ακτίνες. Οπότε, μήπως πρέπει με μια άλλη επισήμανση ή κάτι άλλο, κάποια άλλα στοιχεία στην ε, ταμπέλα να αφήσουμε στην παραγωγή τη συγκεκριμένη αυτή αντιλιακή κρέμα. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Φυσικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή να επιβάλλουμε σε κάποιον παραγωγό αν θα παράγει ή όχι. Αλλά αν θέλουμε να προσφέρουμε ένα πραγματικά φυσικό προϊόν για την προστασία από τον ήλιο, θα πρέπει όντω να δούμε τι γίνεται ε, και με το, με το 1 προ 3 που πρέπει να προστατεύει από τις ακτίνε UVA και UVB. Οπότε, μέσω μιας τέτοιας ε, κρέμας, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει τόση φασαρία, δεν έχω όπλα πάνω μου. Το ερώτημα λοιπόν, η παραγωγή μπορεί να διατηρηθεί, μπορεί να προσφέρεται στο ε, κοινό η κρέμα αυτή αλλάζοντας την επισήμανση. Γιατί φυσικά η προστασία από τον ήλιο είναι πολύ σημαντική, αλλά βέβαια πρέπει να δούμε και το θέμα της ε, ανεκτικότητας από το δέρμα. Jeg øh, sige, at jeg synes, det er meget, det er meget vanskeligt for os at Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι για μας είναι δύσκολο να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε μια θέση και να πούμε κατά πόσο ένα προϊόν προκαλεί αλλεργίες ή όχι. Αυτό πρέπει να το εξετάσουν οι επιστήμονες. Εκείνοι θα αποφασίσουν. Υπάρχουν ένα σωρό φυσικά προϊόντα που μερικές φορές είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Όταν λέμε ότι ένα φυσικό προϊόν δεν είναι επικίνδυνο, αυτό δεν είναι ένα επιχείρημα που στέκει. Γιατί μπορεί να είμαστε αλλεργικοί και σε τελώς φυσικά προϊόντα. Γι' αυτό καταλαβαίνω την επιχειρηματολογία της Επιτροπής που λέει ότι δεν αλλάζει τίποτα. Ο παραγωγός μπορεί να στηρίξει το προϊόν του. Δεν είμαστε εμεί που θα αποφανθούμε για το κατά πόσο είναι επικίνδυνο ή δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε έτσι εξορισμού ότι κάθε φυσικό προϊόν δεν είναι επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να υπάρξει τοξικότητα από ένα φυσικό προϊόν. Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω σε διάφορα σημεία που ακούστηκαν. Υπάρχει η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είπαμε, και υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται από τον κλάδο προκειμένου να βελτιωθεί η σήμανση των ε, προϊόντων αυτών, των καλλιντικών, λαμβάνοντα υπόψη τη σύσταση. Στη νέα σήμανση λοιπόν, η βιομηχανία καλλιντικών κατέληξε σε ένα σήμα που δηλώνει την προστασία από τις υπεριόδιες ακτίνες με νούμερο 1, 2, 3. Υπάρχει ένα μίνιμουμ λοιπόν που προστατεύεται το δέρμα από την ακτινοβολία αυτή. Έγινε μια πρόταση που έλεγε ότι τα φυσικά προϊόντα τα οποία δεν τηρούν αυτό το ελάχιστο ποσοστό να μην χρησιμοποιούν το σήμα. Αυτό θα ήταν μια λύση. Υπάρχει ένα σχόλιο τώρα και για τα φυσικά προϊόντα. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι και τα φυσικά προϊόντα μπορεί να προκαλούν αλλεργίες. Γι' αυτό και δεν συμφωνούμε με την άποψη της βιομηχανίας που λέει ότι τα εντελώς φυσικά προϊόντα δεν προκαλούν αλλεργίες ή δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουν εξανθήματα, γιατί μερικές φορές μπορεί. Αυτά είναι τα κυρία σημεία που ήθελα να αναφέρω. Μπορούμε να ζητήσουμε από τον παραγωγό να μην χρησιμοποιεί αυτό το σήμα, να αλλάξει σήμα και να μεταφέρει προς τους καταναλωτές διαφορετικά το γεγονός ότι το, προστατεύει το δέρμα σε ένα βαθμό η κρέμα αυτή. Χωρίς όμως να προστατεύει εξίσου όπως και οι εντυλιακές εκείνες κρέμες που φέρουν το σήμα προστασίας από τις υπεριόδες. Πρέπει να δούμε πώς η παραγωγή θα ε, διασφαλίσουν επίσης τον τρόπο παραγωγής των συστατικών, κατά πόσο είναι εντελώς φυσικός ή όχι. Γιατί αυτό το διοξείδιο μπορεί να προκαλέσει χημικές αντιδράσεις. Για να έχουμε το διοξείδιο του τανίου δηλαδή χρειάζεται μια χημική αντίδραση. Οπότε είναι δύσκολο να μιλήσουμε για καθαρά ε, φυσικό προϊόν τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς περνάει από μια χημική αντίδραση. Είναι αναγκαίο για να έχουμε αντιλιακή κρέμα. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν η πρόταση του να ζητήσουμε μια περαιτέρω γνωμοδότηση από πλευρά τη Κομισιόν για την εσωτερική αγορά Μπορεί να σας βρει σύμφωνος για να έχουμε περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση για το πρόβλημα της ετικετοθεσίας για την αναγραφή δηλαδή των στοιχείων για το προϊόν, των συστατικών μάλλον του προϊόντος. Μπορούμε να ζητήσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις αν συμφωνείτε. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Το ερώτημά μου ήταν το εξή. Ε, υπάρχει η συγκεκριμένη διάταξη. Δύο λεπτά να αλλάξω και μικρόφωνο. Οπότε πρέπει να υπάρχουν κάποιε προποθέσει που να πληρούνται. Ένα, ένα προ τρία δηλαδή μεταξύ UVA και UVB. Οπότε κανεί μπορεί να περιγράψει μια κρέμα ω αντιλιακή κρέμα, αν πληρεί αυτέ τι προποθέσει. Αν τώρα δεν μπορεί ο παραγωγό να, το παρα... να ε, εγγυηθεί αυτή τη σχέση ενό προ τρία, τότε δεν μπορεί να θεωρήσει την κρέμα αυτή ω αντιλιακή. Μπορεί να, την, ε, να συνεχίσει όμως να την προσφέρει, να την, ε, να την δίνει στην αγορά. Μπορεί να πει ότι ναι, εν μέρη προστατεύει, αλλά να έχει μια διαφορετική επισήμανση αυτή η κρέμα που δεν θα θεωρείται πια αντιλιακή. Αυτό είπα εγώ. Ίσως ο παραγωγός να πρέπει να ζητήσει να γίνει αυτή η αλλαγή. Γιατί έτσι δεν θα μείνει και κανένα α, θέμα εκρεμές. Οπότε γίνεται η παραγωγή, μπαίνει η επισήμανση, ε, εφόσον θέλουμε, αν μπορούμε να αλλάξουμε την επισήμανση, τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι τι λένε. E Η παραγωγό που εκπροσωπεί την εταιρεία έχει κάτι να προσθέσει. Ε, προσπάθησα να, είναι, να είμαι σαφής γιατί δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν και υποπτικές αρχές και στο παρελθόν είδαμε ότι τέτοιες ε, συστάσεις κάποια στιγμή γίνονται οδηγία, ε, μπαίνουν σε μια οδηγία. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε πολλές ε, ευκαιρίες, δεν θα έχουμε πολλές δυνατότητες για να είμαστε επιτυχείς. Τώρα αν θα είναι φυσικό, μη φυσικό, χημικό το φίλτρο για την προστασία από τον ήλιο, δεν είναι αυτό ζωτική σημασία. Ζωτική σημασία είναι να μην έχουν αυτά τα ε, προϊόντα διοξίτη του τιτανίου. Υπάρχουν πολλοί καταναλωτές και πολλοί αλλεργικοί καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα φυσικά προϊόντα που χρησιμοποιούν και έχουν και καλή εμπειρία με αυτά τα προϊόντα. Ας πούμε, οι αλλεργικές αντιδράσεις στα... ή η πρόκληση τέτοιων, η πρόκληση ασθενειών από ε, καλλιτικά που έχουν φυσικά μέσα προστασίας. Ποια είναι, μπορούμε να τη μάθουμε κάπως. Δεν αλλάζει η θέση γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση. ως συνέπεια της σύστασης στην αγορά. Θα αρκούσε μια προσθήκη στο σήμα, στην ε, ετικέτα. Θα πρέπει ο καταναλωτής να διαπιστώνει σε τι βαθμό προστατεύει το προϊόν, τι επιπτώσεις προκαλεί ακόμα και αν δεν αναγνωρίζεται αυτό επίσημα. Οπότε, για την ε, αναφορά αυτή θέλουμε παραπάνω διευκρινήσεις ή δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Και υπάρχει κάποια απάντηση από την Επιτροπή μας μετά από την μελέτη που κάναμε σε βάθος που λέει ότι μπορεί κάλλιστα να επανέλθει στην αγορά, στο εμπόριο δηλαδή η κρέμα αυτή αρκεί να αλλάξει η ετικέτα. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα και να ενημερώσουμε τις αναφέρουσες προ αυτή την κατεύθυνση. Καλώς. Ωραία. Κλείνει λοιπόν με την ανακοίνωση αυτή που θα καταλήξει στις αναφέρουσες. Και πάμε στο 6 που είναι 33-2009 του Κλάους Λάνταν, γερμανικής ηθαγένειας. Ήρθε τώρα και εκπρόσωπος Επιτροπής, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Νικολακόπουλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Um, η κυρία Νικολακόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή η αναφορά θίγει το πολύ σημαντικό θέμα της, ε, της και της αναφοράς αυτήν την ετικέτα της προέλευσης και έχουμε μάλιστα καινούργια πρόταση της Κομισιόν για την παροχή πληροφοριών περί τροφίμων προς τους καταναλωτές. Θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ε, ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία η αναφορά της ε, προέλευσης της καταγωγής είναι προαιρετική και απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές μπορεί να παραπλανηθούν όσον αφορά την πραγματική καταγωγή ή προέλευση των τροφίμων. Επίσης είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις ε, ορισμένων τομεακών κανόνων στο πλαίσιο της κάθετης νομοθεσίας, για παράδειγμα για προϊόντα όπως ο ίνος, το ελαιόλαδο, ποροκυπευτικά, μέλι, ε, βόλιο κρέας, ε, εισαγόμενο κρέας πουλερικών και ε, ηχθείς. Παρατηρούμε λοιπόν πως είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τέτοιες πληροφορίες δίνονται να μην είναι παραπλανητικές για τον καταναλωτή θα θέλαμε να βελτιωθεί η ε, νομοθεσία περί επισήμανσης ε, έτσι ώστε οι καταναλωτές να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τα χαρακτηριστικά και τις ε, ιδιότητες των τροφίμων καθώς και τη διατροφική τους σύσταση. Ξετάζουμε στο πλαίσιο της νέας πρότασης για την ενημέρωση περιτροφίμων, τις πληροφορίες μάλλον περιτροφίμων και η διαβούλευση καθώς και η μελέτη αξιολόγησης πριν από τη σύνταξη της πρότασης δεν έδειξαν ότι η επιβολή της επισήμασης της προέλευσης σε κοινοτικό επίπεδο είναι δικαιολογημένη και αυτό διότι η ζήτηση για τις πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή προέλευση ε, ποικίλει από κράτος μέλος σε μέλος και δεν είναι κάτι το οποίο αφορά όλα τα τρόφιμα, αλλά μόνο ορισμένα εξ αυτών. Γι' αυτό η νέα πρόταση διατηρεί την αρχή ότι η επισήμαση περί προέλευσης είναι, είναι προαιρετική και καθίσταται υποχρεωτική μόνο σε περιπτώσεις όπου δύναται να παραπλανηθεί ο καταναλωτής. Ωστόσο, όσον την ε, προαιρετική ενημέρωση για την προέλευση, η νέα πρόταση της Κομισιόν δίνει ε, περισσότερους ε, κανόνες όσον αφορά την μη παραπλανητική ε, φύση των πληροφοριών που δίνονται σε περίπτωση κούσιας ενημέρωσης. Δίνεται το παράδειγμα της Μαρμελάδας όπου λέει ότι αν δίνονται πληροφορίες για τη χώρα ε, προέλευσης ε, σημαίνει πως το προϊόν αυτό έχει παραχθεί στην, χώρα, στην λόγω χώρα και ότι ε, υπέστη και την τελευταία πιο σημαντική μεταπίση στην ίδια χώρα. Ωστόσο, η πρόταση απαιτεί επίσης την υπόδειξη της προέλευσης ή του χώρου προέλευσης των κυρίων συστατικών. Όταν αυτά τα συστατικά προέρχονται από μέρος που είναι διαφορετικό από την ε, καταγωγή του τελικού προϊόντος. Αν για παράδειγμα η μαρμελάδα για την οποία μιλούσαμε λέει ότι είναι μαρμελάδα από την Νότια Αφρική, σημαίνει πως και τα φρούτα είναι από την Νότια Αφρική. Αντιθέτω. αν, ε, αν τα φρούτα προέρχονται από άλλη χώρα, τότε ο, ο, κατασκευαστής θα πρέπει να υποδείξει την προέλευση αυτών των συστατικών. Όλα αυτά στο πλαίσιο της νέας αυτής πρωτοβουλίας που προέρχεται από την ε, ΓΔ Γεωργία και αφορά την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, όπου επίσης το θέμα του, σημείου, του, του χώρου μάλλον καλλιέργειας συζητείται. Οι απαντήσεις είναι αποτέλεσμα μιας πράσινης βίβλου, ενός πράσινου βιβλίου που οι ενδιαφερόμενοι ερωτήθηκαν κατά πόσο η καταγωγή, ο χώρος, ο τόπος παραγωγής, καλλιέργεια θα πρέπει να αναφέρονται και εδώ στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης είχαμε αντιπαρατηθέμενες απόψεις γιατί καταναλωτές και παραγωγοί υποστηρίζουν ε, τις επιπλέον πληροφορίες για το τόπο παραγωγής αλλά οι λιανοπολιτές αλλά και οι πολιτές χονδρικής ε, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου σε σχέση με την υπερβολική παροχή πληροφοριών ε, Η πρόταση λοιπόν για την ενημέρωση για τα τρόφιμα, τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, αλλά και για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων εξετάζονται, είναι υπό εξέλιξη η εξέταση αυτών των δύο προτάσεων και σίγουρα σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε τα τελικά αποτελέσματα αυτής της συζήτησης. Θα σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο που θέλει να πάρει το λόγο? Εγώ πιστεύω ότι αφού άκουσα την απάντηση της Επιτροπής, ε, μπορούμε να πούμε πως εξαντλήσαμε την ερευνά μας γιατί η απάντηση ήταν ε, πολύ εμπεριστατωμένη για τα ερωτήματα που ε, τέθησαν και ίσως θα ήταν σκόπιμο δεδομένες της συζήτηση που έχει ανοίξει στην Επιτροπή Γεωργίας να κλείσουμε αυτή την αναφορά και να διαβιβάσουμε τα πρακτικά μας στην Επιτροπή Γεωργίας αλλά και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς αν συμφωνήσετε και εδώ να κλείσουμε την αναφορά μας. Ωραία, τέλεια. Περνάμε στην στο σημείο μάλλον 8 που αφορά την αναφορά 1428 του 2009 την οποία υπέβαλε ο κύριος Κώστερ που δεν είναι παρόν και θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο, την εκπρόσωπο της Επιτροπής της Ιζάν Χούκερ. Ευχαριστώ. Ζητάει ο αναφέρον να μην γίνονται δοκιμές για καλλιντικά πάνω σε ζώα και να στηρίξουμε προϊόντα, μάρκες που μας διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουν πειραματιστεί πάνω σε ζώα για τα καλλιτικά τους. Υπάρχει νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει για τα τελικά προϊόντα καλλιτικών πειράματα σε ζώα. Από το 2004 και από το 2009 για ε, προϊόντα τα οποία περιέχουν ε, κάτι το οποίο έχει πειραματιστεί πάνω σε ζώα. Και από 11 Μαρτίου θα καλύπτονται και οι περιπτώσεις τοξικότητας. Του χρόνου θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Πιστεύουμε ότι οι ανησυχίες του αναφέροντος αντικατοπτρίζονται στην κοινοτική νομοθεσία ήδη. Θέλει κάνει το λόγο. συνάδελφος ε, πιστεύω πως είναι πραγματικά μια βελτίωση γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό και κατά την άποψή μου το πρόβλημα έχει ως εξής. Οι επιστήμονες προχωρούν πολύ πιο πέρα από τις αρχές ε, έγκρισης ε, όσον αφορά τα υποκατάστατα προϊόντα ή τις διαδικασίες ε, τις εναλλακτικές για τις δοκιμές σε ζώα. Συχνά οι δοκιμές αυτές μπορούν να γίνουν πάνω σε κύτταρα. Το θέμα είναι αν αναγνωρίζονται αυτού του είδους οι δοκιμές. Πρέπει να ενθαρρυνθεί λοιπόν η Κομισιόν στη διαδικασία αναγνώρισης, ε, επιβεβαίωσης των δοκιμών γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην εγκατάλειψη των δοκιμών ε, σε ζώα αν αυτού του είδους οι δοκιμές ε, αναγνωρίζονταν. Δεν είναι θέμα λοιπόν επιστημονικό, δεν είναι θέμα προ... επιστημονικής πρόοδου, είναι θέμα αναγνώρισης, αμοιβαίας αναγνώρισης των δοκιμών αυτών. Θα πρέπει η Κομισιόν λοιπόν να μας πει αν μπορούμε όντως να κάνουμε ένα άλμα σε αυτό το τομέα. θα πρέπει να διερωτηθούμε αν τελικά είναι απλώς μια συνήθεια το να καταφεύγουμε σε δοκιμές σε ζώα ή κατά πόσο η... ο δεν είναι αρκετά καινοτόμο. Εγώ πιστεύω πως μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ πιο μακριά από ό,τι κάνουμε για την ώρα. Υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη σειρά από πράγματα που δεν χρειάζεται να γίνονται πλέον δοκιμές σε ποντίκια ή σε άλλου είδους ζώα. Εγώ ασχολούμαι το θέμα εδώ και 10 χρόνια περίπου και έχουν γίνει πολλές πρόοδοι. Και έπειτα όταν κοιτά κανείς τους αριθμούς στις εκθέσεις διαπιστώνει πως ο αριθμός των δοκιμών στα ζώα αυξάνεται αντί να γίνεται το αντίθετο. Υπάρχουν παραγωγοί που λένε ναι, εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω εναλλακτική διαδικασία, αλλά δεν ε, έχει αναγνωριστεί ακόμα αυτή η διαδικασία. Άρα στην ουσία χρονοτριβούμε. Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να προχωρήσει πιο γρήγορα, πιο μακριά στη διαδικασία αναγνώρισης αυτών των εναλλακτικών δοκιμών. Η συνάδελφος Όκεν. Øh, <clears throat> øh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ στην αρχή της δεκαετίας του 90 ήμουνα για τέσσερα χρόνια μέλος της ε, αρχής που ήταν υπεύθυνη για, τους, ε, για τα πειράματα σε ζώα. Οπότε ε, εκπροσωπούσα, ας πούμε, την πλευρά, την οπτική γωνία των, ε, των ζώων. Και αν κανείς προσπαθήσει ε, να υπερασπιστεί αυτή την οπτική γωνία, αυτό είναι πάρα πολύ δαπανηρό. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τα ζώα για τα οποία θα πρέπει, δεν θα πρέπει να γίνονται, πάνω στα οποία δεν θα πρέπει να γίνονται ε, πειράματα, αλλά μιλούμε και για το, τα, τις δαπάνες που θα επιφέρει αυτό Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα μια καλύτερη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό, στις ε, ΗΠΑ. Αν υπάρχει κάπου ένα πρόβλημα, έρχεται, με ένα, έρχεται ένα αεροπλάνο γεμάτο με δικηγόρους και λύνει το θέμα. Αλλά εμείς εδώ έχουμε το θέμα το ότι ο παραγωγός είναι ο υπεύθυνο. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν αν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για το αν μία ε, δοκιμή σε ζώα επιτρέπεται να γίνει. Γιατί δεν γίνεται να πιστεύουμε απλώς ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιλικοί προς τα ζώα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να νομίζουμε απλώς ότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους ε, καταναλωτές, να προστατεύσουμε και τα ζώα. Ναι μεν, αλλά σημαντικό είναι εδώ να, να δούμε και τα οικονομικά ζητήματα τα οποία μπαίνουν στο παιχνίδι από την πλευρά του παραγωγού. Υπάρχει μια οδηγία, την προετοιμάζαμε 10 χρόνια, η οποία είχε, στόχος, είχε στόχο τα πειράματα να καταργηθούν πλήρως ό,τι αφορά τα καλλιντικά τουλάχιστον. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που άργησα, οπότε δεν άκουσα και όλη τη συζήτηση. Οπότε, αν πω πράγματα που ήδη έχουν υποθεί, συγχωρήστε με. Ε, αυτό που είπε ο κύριος Γιάννη για το ρυθμιστικό, τις ρυθμιστικές δομές που μπορούν ίσως να αποτρέψουν τους ερευνητές και τους παραγωγούς για να, από τη χρήση τέτοιων μεθόδων πειραματισμού σε ζώα. Αν αυτό συμβαίνει, τότε πρέπει κάτι να γίνει. Νομίζω ότι όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο θέλουμε να αποφεύγουμε τέτοια πειράματα σε ζώα που είναι ζωντανά, εάν αυτό είναι δυνατό να γίνει. Οπότε θα ήθελα με μεγάλο ενδιαφέρον να μας πει η Κομισιόν την άποψή της. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί. Και αυτό που είπε η κυρία Όκεν επίση είναι σημαντικό για το κόστος των δοκιμών σε ζώα. Συχνά υπάρχει αυτή η ιδέα όσων ε, ε, διαδηλώνουν εναντίον των, ε, των πειραμάτων αυτών που λένε ότι είναι πολύ κακοί οι επιστήμονες που θέλουν να τυραννούν τα ζώα. Ε, αυτό είναι λάθος. Ούτε οι ερευνητές θέλουν να τυραννούν τα ζώα και φυσικά είναι και πάρα πολύ δαπανηρή όλη η διαδικασία και πάρα πολύ ε, στεγανή και πολλοί θα ήθελαν να έχουν αναλλακτική λύση για τα πειράματα αυτά. Και επίσης κυρία Πρόεδρε, σήμερα το πρωί στα ΜΜΕ ακούστηκε κάτι για ένα νέο ε, εμβόλιο που υπάρχει για, τον, ε, για την αντιμετώπιση του ε, καρκίνου του στήθους, του καρκίνου του μαστού ποντίκια χρησιμοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα ήταν πολύ επιτυχή. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς γίνεται το πείραμα, εκτός αν κάνεις το πείραμα σε όλο το ζώο και όσοι θέλουν να καταργήσουν ε, πλήρως τα πειράματα σε ζώα. Ε, εγώ εκπροσωπώ 4,2 εκατομμύρια άτομα. 2,1 εκατομμύρια είναι ε, γυναίκες. Ε, οπότε δεν μπορώ να τους πω, να πάω πίσω και να τους πω ότι εμείς καταργήσαμε τα ε, εμβόλια για, αυτό το συγκεκριμένο, ε, για αυτή τη συγκεκριμένη πάθηση μόνο και μόνο για να σώσουμε τη ζωή 12 ποντικιών. Ευχαριστώ. No, Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ναι, ο κύριος Μποστινάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η προσέγγιση είναι αρκετά επιστημονική και τεχνική και μπορεί εμείς εδώ να ε, χρωματίσουμε τη συζήτηση με, με πολιτικό πάθος και να μην καταφέρουμε να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως και ο συνάδελφος Γιάρα, αυτές τις δοκιμές και αξιολογήσεις και να θυμίσω ακόμη στους συναδέλφους που ήταν στην αντιπροσωπεία στην Ισπανία ότι είπαμε το ίδιο πράγμα, ότι υπάρχουν δηλαδή κάποιες, κάποιες έρευνες που αναφέρονται σε ραδιοενέργεια ή δοκιμές σε ζώα ή σε ε, κύτταρα υπάρχουν ορισμένα δοκιμ... ορισμένες δοκιμές ή πειράματα που δεν αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάθε ε, μέρος ε, αμφισβητεί την ε, σοβαρότητα του άλλου μέρους και του δικού του πειράματος και εξ αυτού προκύπτουν ε, διαφωνίες. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεχόταν ένα στόχο του να προχωρήσει προς την οικονομική διακυβέρνηση και να αξιολογήσει τα εθνικά πειράματα πριν να φτάνουν στις εθνικές ε, βουλές, νομίζω πως θα μπορούσαμε και να εισάγουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό για την αναγνώριση των εργαστηριακών ε, δοκιμών. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό. ώστε να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στην επιστήμη να εξελιχθεί, να προχωρήσει και ταυτόχρονα να μειώσουμε τον αριθμό πειραμάτων σε ζώα. Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην μπορεί να φτιάξει μια νομική βάση, μια θεσμική βάση μέσω της οποίας ορισμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια να πιστοποιηθούν ώστε να μπορούν να εγκρίνουν ορισμένες ε, δοκιμές. Η χρήση ζώων και τα πειράματα σε ζωντανά ζωά στα καλλιτικά ή στα φάρμακα σχετίζεται με την φύση του θέματος, του αντικειμένου. Και πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναζητήσει μια ευρωπαϊκή λύση για αυτού του είδους τις δοκιμές. Μια ευρωπαϊκή αναγνώριση για αυτού του είδους τις δοκιμές που αργότερα θα επιτρέψουν και την επιστημονική πρόοδο που θα οδηγήσει στην μείωση των πειραμάτων σε ζωντανά ζώα. Ευχαριστώ. Δεν ζητά κανεί άλλο το λόγο. Η υπεύθυνο τη Επιτροπή δεν ξέρω αν έχει κάτι παραπάνω να μα πει. Θέλει κάτι να προσθέσει, μάλιστα. Για να δούμε το θέμα από την άποψη των καλλιτικών. Υπάρχει μια πολιτική απόφαση που έχει ληφθεί μέσω της οδηγίας ε, για τα καλλιτικά. Πρόκειται για πλήρη απαγόρευση άσχετα από το κόστος ή τη διαθεσιμότητα των μεθόδων. Ε, ε, αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε. Ήδη έχει ληφθεί η απόφαση αυτή και έχει γίνει η επιλογή. Τώρα για να εξετάσουμε την επιστημονική διαθεσιμότητα διαφόρων μεθόδων αυτό θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την οδηγία των καλλιτικών πριν μετά από το Μάρτιο του 2011 γιατί ούτως ή άλλως ε, οι κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία μέσω μιας πολύ περίπλοκης διαδικασίας και έχουμε αρχίσει την ε, σχετική εργασία μαζί με το Κοινό Κέντρο Ερευνών και με διάφορους εμπειρογνώμους για να δούμε πού βρισκόμαστε. Η εντύπωσή μας είναι ότι δεν είμαστε ακόμα σε, κοντά στην έγκριση τέτοιων ε, δοκιμών, εναλλακτικών δοκιμών, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας ενημερώνουμε στο Κοινοβούλιο για το πού βρισκόμαστε. Και όσον αφορά την επικύρωση των μεθόδων, το Κοινό Κέντρο Ερευνών έχει καθιερωμένο τρόπο, θεσπισμένο τρόπο για την αξιολόγηση των εναλλακτικών μεθόδων και έχουν γίνει προσπάθειες για την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας, αλλά για το θέμα της ε, οδηγίας για τα καλλιτικά δεν υπάρχουν αυτές οι μέθοδοι. Δεν έχει να κάνει με την επικύρωση αυτών. Δεν υπάρχουν εναλλακτικέ μέθοδοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα που σίγουρα ε, μας βρίσκει όλους σύμφωνους όσον αφορά την αντίθεσή μας στην χρήση ζώων για γενικά πειράματα. Εγώ θα πρότεινα να κάνουμε μία παύση για να προβληματιστούμε για το θέμα αυτό, γιατί έχουμε τις επόμενες έξι ε, αναφορές που αφορούν αυτό το ίδιο θέμα, δηλαδή γενικότερα το θέμα των πειραμάτων επιζών για την παραγωγή. Ίσως λοιπόν να ακούσουμε και τις άλλες, ε, τους άλλους προβληματισμούς, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα και να αποφασίσουμε στο τέλος, αφού θα έχουμε ακούσει και την παρέμβαση της Κομισιόν για τις υπόλοιπες έξι αναφορές. Να περάσουμε και να εξετάσουμε την 9 τώρα, την αυτή που είναι στο σημείο 9, 115 του 2008, την 252 2008, 805 του 2009. Να δώσουμε το λόγο στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, Σουζάνα Λούμες. Uh, uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε με την άδειά σα, θα ήθελα να συμπεριλάβω και το σημείο 10, μια που οι δύο αυτέ αναφορές έχουν το ίδιο αντικείμενο. Όλες αυτές οι αναφορές λοιπόν έχουν άμεση σχέση με την οδηγία 8669 όσον αφορά την χρήση πειραματόζων για επιστημονικούς σκοπούς. Επιπλέον λοιπόν από την πρόσφατη απάντησή μας. Θα ήθελα την γραπτή, θα ήθελα και προφορικά να σας μιλήσω για τις εξελίξεις όσον αφορά την μεταρρύθμιση, την, αναρρύθμι, την αναθεώρηση της οδηγίας αυτής και τη συνέχεια. Υπάρχει πολιτική συμφωνία επί της ουσίας που το Δεκέμβριο μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Υποσουδικής Προεδρίας και στην τελική συνεδρίαση της 7ης Απριλίου υπήρξε συμφωνία όσον αφορά τα κρεμούντα ζητήματα για την επιτροπολογία, επειδή ξεκίνησε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εδώ πετυχαίνουμε μια ισορροπία με ανάμεσα στην προστασία των ζώων και από την άλλη μεριά ε, την ε, βοήθεια προς ε, την βιομηχανία για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής. Η νομοθεσία λοιπόν, το σχέδιο κειμένου που θα εγκριθεί τελικά πιστεύουμε, έχει τα τρία στοιχεία που ζητάμε. Όσον αφορά το περιεχόμενο και ειδικά για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις αναφορές αυτές, ας κοιτάξουμε. Έχουμε της κυρίας Έρντ για την απαγόρευση πειραμάτων σε μεγάλα ανθρωποειδή. Υπάρχει μια άλλη από τον δόκτωρα που ζητάει να σταματήσουν τα πειράματα σε ζώα και αν υπάρξουν αναλλακτικέ ε, δυνατότητες και υπάρχει το θέμα της απαγόρευσης και από την κυρία Χέμιγουέι που μιλάει εκ μέρου του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Η δέκα τώρα έχει να κάνει με την απαγόρευση της χρήσης κοιλιών και κουταβιών της ράτσας Μπίγκλε για διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα και ζητά διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει να πει ότι το κείμενο πάνω στο οποίο υπάρχει συμφωνία, ε, το κείμενο αυτό καλύπτει όλα αυτά τα θέματα. Θα ζητάει συστηματική ηθική αξιολόγηση. Οπότε άλλη είναι η αισθητική πλευρά και άλλη είναι αυτή η ηθική. Επίσης μιλάει για άδειε που θα πρέπει εκ των προτέρων ε, να έχουν εγκριθεί για να γίνονται πειράματα σε ζώα. Παρακολουθούμε όλο το ιστορικό, όλες τις επιθεωρήσεις, γίνεται και αξιολόγηση εκ των υστέρων. Οπότε, πολλά από τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρωποειδή θα ισχύουν. Υπάρχει απαγόρευση για την χρήση ανθρωπιδών που ζητάνε πολύ από τους αναφέροντες, αλλά υπάρχουν και εξαιρεσει εφόσον υπάρξει ξέσπασμα ασθένειας επιδημίας. Όσον αφορά εναλλακτικέ μεθόδους τώρα, που και αυτό είναι ένα ζήτημα στον τομέα των καλλιντικών, γίνονται πολλοί προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στις απαντήσεις μας το έχουμε συμπεριλάβει, ότι θέλουμε δηλαδή να ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα πλαίσιο, τον έφερε και συνάδελφος πριν, αλλά επιταχύνουμε επίσης και το ρυθμιστικό πλαίσιο σύμφωνα με τόσα ζήτησε ένας ευρωβουλευτής εδώ για εναλλακτικά πειράματα. Το κείμενο όμως καλύπτει τέσσερα σημεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν για να έχουμε καλύτερες μεθόδους πειραμάτων στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα από τα κράτη-μέλη να εντοπίζουν και να ορίζουν ειδικά εργαστήρια ώστε να έχουμε καλύτερη συμμετοχή στην αξιολόγηση. Δεύτερον, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν εναλλακτικέ λύσεις σε εθνικό επίπεδο. Το ίδιο βέβαια ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το διεθνή χώρο. Τώρα στο θέμα της αποδοχής των ρυθμίσεων, είναι εδώ θέμα χρόνου, πόσο καιρό χρειάζεται για να σωματωθεί στην νομοθεσία. Είναι επίση θέμα το πόσο κατάλληλη είναι μία μέθοδο βάσει των ρυθμιστικών απαιτήσεων. Πάντω, η οδηγία θεσπίζεται από το κάθε κράτο μέλο να ορίζει ένα σημείο επαφή ενιαίο όταν πρόκειται για θέματα που έχουν να κάνουν με ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να επιταχυνθεί το έργο και να διευκολυνθεί η δουλειά των υπαλλήλων. Τέλος, ζητούμε από τα ευρωπαϊκά εργαστήρια να φροντίσουν να υπάρξουν εναλλακτικέ μέθοδοι. Μέχρι τώρα δεν υπήρξαν νομική βάση, τώρα λοιπόν δίνουμε νομική βάση σε τέτοιες εργασίες. Και για τα δύο τελευταία, η διαφάνεια ήταν ένα που αναφέρεται κυρίως ε, στην αναφορά που είναι στο σημείο 10. Και έτσι λοιπόν, για τη διαφάνεια, μαζί με την ηθική αξιολόγηση που θα είναι συστηματική, ζητάμε να είναι και αμερόληπτη, και να διέπεται από διαφάνεια. Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται και εκ των υστέρων αξιολόγηση και τέλος αναφορές στατιστικές για την σοβαρότητα των πειραμάτων. Ένα άλλο στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η θέση σε ισχύ η εφαρμογή. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει, πρέπει να γίνεται σωστά. Εμείς πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της διαφάνειας που γίνεται με τα μέτρα αυτά θα βοηθήσει και για την καλύτερη εφαρμογή των μέτρων. Βέβαια, δεν θα πρέπει να εφησυχαζόμαστε και να πιστεύουμε ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται από μόνα τους. Δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρχει και έλεγχος κάθε φορά που υπάρχει κάποια υπόνοια για μη τήρηση των κανόνων, ώστε να μπορούν επιθεωρητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνουν και να ελέγχουν επιτόπου. Τώρα, στη σημερινή διαδικασία, το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει την κοινή του θέση αυτή την ε, εβδομάδα, 3 Ιουνίου, και μετά θα υπάρξει ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο. Τον Ιούλιο στην ε, Επιτροπή και Ολομέλεια το Σεπτέμβριο θα ψηφίσει. Άρα θα αρχίσει να ισχύει και θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο το μέτρο αυτό. Μετά χρειάζονται και μήνες για την εφαρμογή, για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία. Το κείμενο που υποβάλλεται για έγκριση στο Συμβούλιο ε, περιλαμβάνεται σε μια ιστοσελίδα της οποία τα στοιχεία θα αφήσω στη γραμματεία εφόσον θέλετε να μπορείτε να ενημερωθείτε κατευθείαν. Εγώ πιστεύω πως αυτή η παρέμβαση της Κομισιόν έχει δώσει απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που είχαν τεθεί και στην προηγούμενη μας ε, αναφορά. Έχει άρει όλες τις αμφιβολίες. Πιστεύω πως τώρα γνωρίζουμε πως η Κομισιόν έχει πλήρη συνείδηση των ερωτημάτων που έχουμε θέσει. Ένα πακέτο πρωτοβουλειών ε, έχει προετοιμαστεί για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσει και για τη χρήση των ζώων για αυτά τα πειράματα. Θεωρούμε λοιπόν πως αυτή η αναφορά μπορεί να κλείσει και να μεταβάσουμε αυτές τις απαντήσεις στους αναφέροντες των έξι αναφορών. Περνάμε στην αναφορά στο σημείο 11, 12.74.2009 2009 που έχει υποβληθεί από τη Ράκελ Μούλεν. Είναι παρόν, παρούσα ή αναφέρουσα. Δίνω το λόγο λοιπόν στη Ράκελ Μούλεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δουλεύω με, την Alliance. με την Equality Alliance ε, η οποία δουλεύει βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις παραβάσεις που γίνονται σε θέματα ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Η συμμαχία αυτή λοιπόν που εκπροσωπώ εγώ ξεκίνησε το 2008 για να διαμαρτυρηθεί για την ε, διάλυση από πλευρά της κυβέρνησης του φορέου μας. Με 140 μέλη, 83 μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνδικάτα, ακαδημαϊκούς και ενεργούς πολίτες, ανησυχούμε πάρα πολύ για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα όσον αφορά για την ε, διάλυση ουσιαστικά των δομών που προστατεύουν την ισότητα και καταπολεμούν την φτώχεια. Επιπλέον την αναφορά αυτή τη στηρίζουν και ευρωβουλευτέ, δηλαδή ο Πρίνσε Ντερόσε, Νέσο Τσίλντερ, Άλαν Κέλλη, Γκέι Μίτσελ, Μέριετ Μακίνε, Τζιμ Χίγγιν, Σιν Κέλλη, Τζο Χίγγιν και Μάριαν Χάρκιν. Τον Οκτώβριο του 2008 ο προπολογισμό τη αρχή αυτή του φορέα αυτό περικόπη κατά 43% από 5,87 εκατομμύρια σε 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Η επικεφαλής ε, παρετήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 ακριβώς διαμαρτυρόμενος για τις περικοπές που επιβλήθηκαν και πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να είναι φιώσιμος ο φορέας από εκεί και πέρα. Στη συνέχεια παρετήθηκαν και άλλα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι περικοπές αυτές ε, οδήγησαν, ε, συνοδεύτηκαν και από άλλες περικοπές που έγιναν σε διάφορα μέτρα που βοηθούσαν το φορέα μας. Για παράδειγμα, ε, ο προπολογισμό περικόπηκε από 31% τη της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η Συμβουλευτική Επιτροπή επίσης είδε το δικό της προπολογισμό να περιορίζεται 100% και έκλεισε βέβαια φυσικά το Δεκέμβριο του 2008 και άλλη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα είδε τον δικό της προπολογισμό να πέφτει κατά 25% από 1,31 εκατομμύρια σε 0,98 εκατομμύρια. Μιλάτε πιο αργά, λέει η Πρόεδρος. Αυτές οι περικοπές ε, λοιπόν και που έγιναν στους φορείς που στηρίζουν την καταπολέμηση των διακρίσεων και υποστηρίζουν την ισότητα ήταν πολύ δυσανάλογε σε σχέση με άλλε περικοπέ που έγιναν στη δικαιοσύνη ή σε μεταρρυθμίσει νομοθετικέ κλπ. Το 2009 λοιπόν ε, ζητήσαμε έρευνα όσον αφορά τις περικοπές αυτές που επέβαλε η κυβέρνηση στις δομές μας. Η έρευνα αυτή δημοσιεύθηκε αφού ξεκίνησε η αναφορά που βάλαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σημειώνεται εξή ότι η περικοπή του προπολογισμού 43% του φορέα και η μείωση του προσωπικού από 53% σε 38% σημαίνει ότι τίθεται σε αφισβήτηση η δυνατότητα του φορέα να φέρει σε πέρα στο έργο του. Η ανεξαρτησία επίσης του φορέα πλήττεται επειδή δεν υπάρχει αρκετή πρικοδότηση. Το προσωπικό επίσης μειώθηκε, πράγμα το οποίο μας οδηγεί να γινόμαστε υπόλογοι περισσότερο στην κυβέρνηση παρά στο κοινοβούλιο. Η τρέχουσα λειτουργία πάντως της αρχής δεν είναι σε θέση να ε, διαπιστώσει ότι τηρούνται οι αρχές των ε, Παρισίων ή οι συστάσεις της ε, οδηγίας του 2000 RACE. Επιπλέον, το προφίλ του φορεαυτού μειώθηκε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξετάσει τον ίδιο αριθμό περιπτώσεων όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θα ήθελα να επιτρέψω στον συναδελφό μου Όρλε Κοφάρελ να μιλήσει για την νομική βάση, βάση της οποίας καταθέσαμε και την αναφορά αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Όρλε Κοφάρελ. Είμαι ε, ανεξάρτητος φορέας σε θέματα διακρίσεων και παλιά δούλευα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι καταγγελίες μας έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση κάνοντας ε, γενικά περικοπές πλήττει ιδιαίτερα τον ε, φορέα Equality της Ιρλανδίας με δυσανάλογες περικοπές. Οι περικοπές αυτές μαζί με την, το πρόγραμμα αποκέντρωσης που έγινε πάρα πολύ γρήγορα όσον αφορά την περίπτωση του φορέα αυτού υπονόμευσαν την ε, δυνατότητα του φορέα να λειτουργήσει ω σώμα ειδικό για την καταπολέμηση των διακρίσεων και να φέρει σε πέρα τα καθήκοντά του που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Υπάρχει δυσανάλογη επίθεση λοιπόν στο φορέα αυτό σε σχέση με άλλους και πιστεύουμε ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση ουσιαστικά πέρασε από μια κατάσταση που συμμορφωνόταν με το κοινοτικό δίκαιο σε μια κατάσταση που δεν συμμορφώνεται με το κοινοτικό δίκαιο. Βάσει τη κοινοτική νομοθεσία, λοιπόν η αρχή για την ισότητα πρέπει να μπορεί να φέρει σε πέρας ε, πέντε καθήκοντα. Πρώτα απ' όλα να βοηθάει τα θύματα διακρίσεων, ε, υποβάλλοντα καταγγελίε κλπ. Δεύτερον, να κάνει αναλύσει για τι διακρίσεις. Τρίτον, να δημοσιεύει εκθέσεις και συστάσεις. Να προχωράει σε δικαστικές ε, διώξεις στο όνομα των θυμάτων. Και τέλος, πρέπει να είναι ένα ανεξάρτητο όργανο. Τον Οκτώβριο, τον ε, Οκτώβριο λοιπόν του 2008 ο προπολογισμό, όπως είπαμε ε, περικόπη κατά 43% από 5,87 εκατομμύρια σε 3,3 εκατομμύρια. Συγχρόνως υπήρξε αποκέντρωση του φορέα και πήγε σε ένα μακρινό μέρος από το Δουβλίνο και το προσωπικό επίσης ε, κόπηκε στα δύο. Περιορίστηκε το προσωπικό από 53 σε 38 άτομα που σημαίνει ότι χάθηκαν πολλοί άνθρωποι που δούλευαν εκεί με μεγάλη εμπειρία. Τον Αύγουστο του 2009 επίσης παρετήθηκε ο νομικός σύμβουλος ε, του Φορέα και δεν αντικαταστάθηκε. Κάτι το οποίο έπληξε την αποτελεσματικότητα του Φορέα που δεν μπορεί πλέον να φέρει σε πέρα στα καθήκοντά του βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2007 η Επιτροπή έκανε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέγοντας ότι η δυνατότητα ενός σώματος για την ισότητα να λειτουργεί εξαρτάται από τη χρηματοδότησή του. Και επιπλέον το 2007, στο τέλος του Ευρωπαϊκού Έτους ε, Ίσων Ευκαιριών για Όλους, το Συμβούλιο Υπουργών ε, ετοίμασε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε από τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ειδικών φορέων για την ισότητα, ενισχύοντας την ανεξαρτησία τους και προσφέροντάς τους ε, παρά τους Δημοσιονομικού περιορισμού, στου κατάλληλου πόρου. Όμως η Ιρλανδική κυβέρνηση αντί να κάνει αυτό διάλεξε τον φορέα αυτό τον ειδικό για την ισότητα για να κάνει περικοπές στον προπολογισμό πολύ δυσανάλογε με τις περικοπές που έγιναν σε άλλους τομεί. Η Συμμαχία Equality και Δικαιώματα, Ισότητα και Δικαιώματα Διαμαρτύρεται λοιπόν για την περικοπή 43% του προπολογισμού, αλλά και για το γεγονό ότι ο φορέα δεν μπορεί να είναι πλέον αποτελεσματικό. Ο αριθμό των υποθέσεων που άνοιξαν και εξετάστηκαν από τον φορέα έχει περιοριστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Από τότε που έγιναν οι περικοπές δηλαδή. Το θέμα της ανεξαρτησίας είναι ζωτική σημασία γιατί η έρευνα που έγινε από την Ήρα τονίζει ότι πλήττεται η ανεξαρτησία του φορέα και πιστεύουμε ότι ο φορέας της ισότητας τελικά καταδικάζεται, πράγμα το οποίο δείχνει πόσο σοβαρά έχει φροντίσει για την ανεξαρτησία του τομέα αυτού η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Ίσως βέβαια να μην άρεσε στην κυβέρνηση η συμπεριφορά του φορέα που σε πολλές περιπτώσεις έχει καταγγείλει ε, κυβερνητικούς φορείς για τη συμπεριφορά τους. Είτε επειδή κατέγγειλε αξιωματούχους, είτε κυβερνητικούς φορείς. Η αναφορά μας αυτή έχει να κάνει με τις υποχρώσεις που έχει ένα κράτος απέναντι σε έναν φορέα ισότητας. Και εδώ καταγγέλουμε το γεγονός ότι έγιναν δυσανάλογες περικοπές στον προπολογισμό. Εμείς βασιζόμαστε σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίζουν πώ θα εφαρμόζουν ακριβώ τι οδηγίε Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που μπορούν για να είναι αποτελεσματικέ οι οδηγίε και ώστε η εφαρμογή μια οδηγία να μην γίνεται μια και έξω, αλλά να αποτελεί μια συνεχή διαδικασία η οποία υποχρώνει τα κράτη-μέλη να φροντίζουν συνεχώ για την εφαρμογή αυτή και ότι προοδευτικά και σε συνεχόμενα στάδια πρέπει να φροντίζουν για την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών τα κράτη-μέλη. Άρα θα πρέπει να ενισχύεται ένα σώμα για την ισότητα. Εδώ όμως και παρά την απέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ένα ανεξάρτητο σώμα με κατάλληλη χρηματοδότηση για την προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, εδώ αυτό δεν έχει γίνει. Εδώ ανάποδα έχουν πέσει οι προδιαγραφές όσον αφορά τον φορέα ισότητας και άρα έχει καταδικαστεί ο φορέας όσον αφορά το μέλλον του. Έτσι, πλήττεται η αρχή που λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόοδος όσον αφορά την στήριξη της ισότητας από τους εθνικούς φορείς, γιατί αντίθετα εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ε, χαμηλότερο επίπεδο αποτελεσμάτων. Εμείς πήραμε κοινοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία επί παραβάση βάσει των καταγγελιών μας. Και για ποιο λόγο, διότι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό μιλάνε για κατώτερα επίπεδα και άρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Επίσης λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν είναι πεπισμένη ότι η τρέχουσα πρικοδότηση του φορέα αποτελεί εμπόδιο για ε, το έργο της, ε, του φορέα αυτού. Ποιο είναι το επίπεδο. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί μια οδηγία να πει τι επίπεδο πρικοδότησης πρέπει να υπάρχει. Αυτό εξαρτάται στο κάτω-κάτω και από τον πληθυσμό που έχει κάθε χώρα. Όμω η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λέει ότι τα σώματα τα οποία ορίζονται από τι οδηγίε αυτή πρέπει να είναι και ανεξάρτητα αλλά και να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρα αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Έτσι λοιπόν, η... ο φορέα για την ισότητα, δεδομένου ότι μειώθηκε κατά 50% σχεδόν ο προπολογισμό του και περιορίστηκε το προσωπικό κατά 25%, προφανώ και δεν είναι σε θέση να φέρει καλά τα καθήκοντά του σε πέρα. Γι' αυτό και θελήσαμε να έρθουμε εδώ. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να εξετάσετε την αναφορά μας πολύ σοβαρά και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή από μόνη της κάνει έρευνες και στις 27 χώρες για να δει ποια είναι η απόδοση των φορέων για την ισότητα στα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι η αναφορά μας και η καταγγελία μας είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί πολύ υπόψη στα πλαίσια της έρευνας αυτής και δεδομένου ότι υπάρχει και νέα οδηγία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μιλάει για την ανεξαρτησία και την κατάλληλη πρικοδότηση φορέων ισότητας στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Yes, thank you. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ανέκαθεν είχε καλό διάλογο η Κομισιόν με τον αναφέροντα την ε, Συμμαχία Ισότητας και Δικαιωμάτων και Θεωρούμε πάρα πολύ, εξετάζουμε πολύ σοβαρά την, την αναφορά σας. Έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες, έχουμε μελετήσει την ανεξάρτητη μελέτη που εσείς κάνατε ε, και γνωρίζουμε πως όλα αυτά επηρεάζουν ένα μεγάλο κομμάτι της ε, κοινωνίας των πολιτών στην Ιρλανδία. Μόνο δεν μου αφήσατε και πολλά να πω στην ουσία γιατί έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Απλώς να θυμίσω πως ε, τα σώματα ισότητας απαιτούνται από την έκθεση, από την οδηγία η που ασχολείται με την, την ισότητα των φύλων και έχει φτιαχτεί ώστε να προωθήσει την ισότητα αντιμετώπισης και μεταχείρισης και η Κομισιόν ασκεί τις υποχρεώσεις της. Αυτό έχει υπογραμμιστεί, έχει ε, προσφέρει ανεξάρτητη βοήθεια στα θύματα, ανεξάρτητες μελέτες και εκθέσεις, δημοσιεύει καθώς και ξεκινά δικαστικές διαδικασίες εξ των θυμάτων. Στην Ιρλανδία ανέκαθεν ήμασταν μοντέλο καλής πρακτικής, είμαστε καλό παράδειγμα και για άλλα κράτη-μέλη. Φυσικά η Κομισιόν ε, θέλει να λάβει την καταγγελία παράλληλα με αυτήν την αφορά. Το λάβαμε το Σεπτέμβριο του 2009 και η απάντησή μας ήταν ότι οι οδηγίες είναι οι οδηγίες για ελάχιστες προδιαγραφές και δεν διευκρινίζονται επίπεδα. Σε απάντηση σε αυτό, η Συμμαχία Ισότητας και Δικαιωμάτων, απογοητευμένη από την απάντησή μας, είπαν ότι το πραγματικό αντίπτυπος αυτών των πολύ μεγάλων περικοπών θα, γίνουν, θα γίνει εμφανής από το 2010 και μετά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παρά αυτό που φαίνεται να είναι πολλές ε, μαρτυρίες και αποδείξεις από νομικής άποψης δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι θα μπορούσαμε να πάμε στο δικαστήριο και να κατηγορήσουμε την Ιρλανδία πως δεν επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να κάνει την, ε, το έργο της όπως ε, ορίζει η οδηγία. Αν και είναι λυπηρό και μας ανησυχεί στην Κομισιόν και ανησυχητικό, θα πρέπει να έχουμε νομικά δεσμευτικές αποδείξεις πως αυτές οι περικοπές καθιστούν αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο τη... για την αρχή ισότητας να ασκήσει το έργο της. Ίσως στο μέλλον αυτό να φανεί. Στο σα ε, ε, όπως σας είπαμε, είπατε και εσείς, μάλλον κάνουμε αυτή τη μελέτη, αλλά μέχρι ότου να έχουμε αυτές τις αποδείξεις, και γράψαμε και πάλι στην ΙΑΡΕΙ e και είπαμε ότι δεν θα ξεκινήσουμε διαδικασία παραβάση αυτή τη στιγμή. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά πως τα κράτη-μέλη δεσμεύονται για να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των οδηγιών και μετά την μεταγραφή τους και φυσικά θα είμαστε ευγνώμονες για οποιαδήποτε ενημέρωση θα μπορούσαμε να έχουμε και στο μέλλον. Ναι, Ευχαριστώ, κυρία Χάρκιν. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την Κομισιόν για την πολύ θετική απάντησή της. Όντως είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι είναι όντω καλή πρακτική η, αυτή που χρησιμοποιείται από την αρμόδια αρχή τη ε, Ιρλανδία και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί και ω υπόδειγμα σε σύγκριση με τα όσα έχουν ήδη συμφεί. Οι συνάδελφοι από τον ΙΑΡΕΙ e ανέφεραν τα πράγματα πολύ διεξοδικά, οπότε δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα άλλο. Ήταν ε, σαφέστατα αυτά που είπαν. Απλώ κάποια σύντομα σχόλια να κάνω. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι μιλήσαμε για την ανεξαρτησία της ε, αρχής ισότητα. Δεν υπάρχει καμία ε, αμφιβολία ότι η ε, εκτελεστική εξουσία αυτής της αρχής ήταν πολύ αποτελεσματική, δεν φοβήθηκαν να χτυπηθούν με το σύστημα και πραγματικά νομίζω ότι πλήρωσαν και το τίμημα. Έτσι έχουν τα πράγματα και γι' αυτό η Κομισιόν τώρα λέει ότι είναι ε, η υπηρεσία αυτή ένα μοντέλο καλής πρακτικής. Σε κάποιο επίπεδο ίσως να, ήταν, να παρά ήταν καλή η πρακτική που ακολουθούσε για κάποιους που ήταν σε θέση είτε να μειώσουν τον, τον προϋπολογισμό της ή να, τις, να την πλήξουν κάπως αλλιώς 43% μείωση του προϋπολογισμού κατά 43% 6 ε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απολυμμένα από 53% ε, σε μείωση του προσωπικού πολλά τα πλήγματα, αλλά μιλούμε για έναν προπολογισμό με μείωση 43%. Δηλαδή, το, αν ήταν 93% η μείωση του προπολογισμού, θα είχε κάποια άλλη θα κάποια διαφορά. Το θέμα δεν είναι ο αριθμό, είναι άλλο. Είναι το, θέμα είναι τι κάνουν αυτέ οι αρχέ, τα 27 κράτη-μέλη, ποιε είναι οι αποδόσει του σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και των προγραμμάτων αυτών. Μόνο αν τις στηρίξουμε θα έχουμε και ανεξαρτησία και, από την, και αυτή που ζητά η Κομισιόν. Και νομίζω ότι οι αναφέρουσες ε, το είπανε πολύ σωστά για το τι γίνεται στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, όπου το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τέτοιοι φορείς να χρηματοδοτούνται επαρκώ. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς εδώ στην ε, αρχή, ε, στην Επιτροπή Αναφορών πρέπει να επιμείνουμε ως προς αυτό και να δούμε ποια είναι τα ευρήματα της Κομισιόν της δικής της έρευνας και μετά να ξαναέρθουμε στο θέμα αυτό. Uh, thanks very much. And, um, Ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ το, τους αναφέροντες για πολύ ξεκάθαρη και συγκεκριμένη παρουσίαση. Είχαμε ασχοληθεί με τέτοια θέματα με τον Επίτροπο Σπίτλα όταν λίγο πριν ε, τελειώσει η θητεία του. Νομίζω πως υπάρχει μια δυναμία στην ισχύουσα οδηγία. Εφόσον η αρχή είναι ότι πρόκειται για μια οδηγία ελάχιστων προδιαγραφών, Ταυτόχρονα η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε όλες οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στην οδηγία να μπορούν να ε, διεξαχθούν. Δηλαδή το αρμόδιο σώμα να μπορεί να ε, ασκεί όλες αυτές τις λειτουργίες. Το θέμα είναι ποιες είναι αυτές που οι λειτουργίε οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να πληρούνται ώστε να πούμε ότι εφαρμόζεται σωστά η έκθεση ή συγγνώμη η οδηγία. Δηλαδή μια έκθεση το χρόνο, ένα πρόγραμμα το χρόνο. Δηλαδή τι θεωρεί μίνιμουμ το ελάχιστο Κομισιόν ή μήπως το αφήνεται σε ό,τι έχει την καλή να χρηματοδοτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει σίγουρα η εν λόγω οργάνωση δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως ε, λειτουργούσε μέχρι τώρα. Έχασε τον νομικό τη σύμβουλο, έχασε ένα μεγάλο κομμάτι του προσωπικού τους, έχει μοιραστεί σε δύο κέντρα, δηλαδή ανάμεσα στο Δουβλίνο και στο Τιπερέρι, σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε προηγουμένως. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κομισιόν επανειλημμένως έχει πει πως η Ιρλανδική Αρχή όπως λειτουργούσε ήταν ένα πρότυπο καλή πρακτική τότε δεν καταλαβαίνω πώς ε, συνδέονται όλα αυτά λογικά. Ε, είναι σαν μια υπόθεση κάτσε 22, δηλαδή ένα διέξοδο. Ωστόσο νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε την οδηγία αυτή Μήπω λοιπόν θα πρέπει και το Συμβούλιο να επαναξετάσει αυτή την οδηγία για να κάνει κάποιες απαραίτητε αλλαγές. Σίγουρα θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η ε, αναφορά αυτή. Αλλά να ζητήσουμε και από την Κομισιόν να φτιάξει κάποιο είδους ε, οριοθέτηση, κάποιο είδους βαθμολόγηση όσον αφορά την τήρηση των ελαχίστων κριτηρίων των ελαχίστων προδιαγραφών. Γνωρίζουμε πω αρκετά κράτη-μέλη έχουν ακολουθήσει την Ιρλανδία όσον αφορά τι περικοπέ στον προπολογισμό. Οπότε μπορεί να γενικευθεί αυτή η οπισθοδρόμηση. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να βρούμε την ισότητα σε ολόκληρη την Ένωση, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης, γιατί είναι στις οδηγίες αυτό αναγεγραμμένο, δηλαδή η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πρόθεση της ισότητας. Πρέπει να μείνει ανοιχτό και πρέπει κάτι να μας φέρει η Κομισιόν σε λίγους μήνες, όχι μόνο σε σχέση με την εξέταση από άλλες αρχές και άλλες κράτη-μέλη, αλλά τι θα πει μήνυμο, ελάχιστο. Σε ποια φάση δηλαδή θα θεωρήσει η Κομισιόν ότι έχει υπάρξει παραβίαση είτε από την Ιρλανδία είτε από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι μήνυμα ανάγκες ε, που θα πρέπει να καλυφθούν και να ξαναεξετάσουμε την οδηγία. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφος Higgins. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν παρουσίασαν την αναφορά του η κυρία Μόλαντ και η κυρία Φάρελ πραγματικά μιλούν εξ ονόματο πολλών στην Ιρλανδία και μιλούν κυρίω για αυτές ε, αυτά τα στρώματα τη ε, Ιρλανδική κοινωνία που χρειάζονται μια φωνή για να ακουστούν ειδικά όταν θέλουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά του στην ισότητα. Οπότε θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που μα είπαν. Όταν ο πρώην εκτελεστικό διευθυντή ε, της ε, αρχής ε, παρετήθηκε λόγω των περικοπών έδωσε μεγάλη, ε, δόθηκε μεγάλη σημασία στην, στο, στη μείωση του 43% και όχι στο 2-3% των περικοπών που έγιναν σε άλλες υπηρεσίες. Οπότε είχε κάτι στο μυαλό της η Ιρλανδική κυβέρνηση. η ισότητα πρέπει να γίνει πράξη κάποια στιγμή. Η απάντηση τώρα της Κομισιόν δεν με πείθει. Αλλά ούτως ή άλλως και η Κομισιόν ε, εδώ πέρα είναι μια, δείχνει από μόνη της και μια μεγάλη αντίθεση. Σε όλη την Ευρώπη προσπαθεί να πιέσει όλες τις κυβερνήσεις για να μειώσουν τις, ε, τα δημοσιονομικά τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους καρχαρίες των χρηματοπιστωτικών αγορών. Κάτι παρόμοιο γίνεται και, στην, και με την Ιρλανδική κυβέρνηση. Για κάθε τέτοιο πρόγραμμα θέτει τέτοια προγράμματα σκληρά, αυστηρά, για να αντιμετωπίσει δίθεν την κρίση. Αλλά όταν η Κομισιόν δεν καταδικάζει την Ιρλανδική κυβέρνηση και επιμένει ότι οι πόροι όντω σε ένα βαθμό πρέπει να δίδονται για την ισότητα. Ε, τότε πώς, τι να περιμένουμε από την Κομισιόν. Η αντίθεση σε αυτό που λέει η Κομισιόν είναι σαφή γιατί λέει από τη μια ότι για να μπορέσουν οι αρχές αυτές σε εθνικό επίπεδο να λειτουργήσουν πρέπει να έχουν επαρκείς πόρους για να μπορέσουν να, να κάνουν όλα τα καθήκοντα που τους έχουν αποδοθεί. Και από την, και την άλλη λέει ότι παρόλα αυτά οι οδηγίες είναι οδηγίες των προτύπων και δεν, και δεν δίνουν συγκεκριμένα επίπεδα ε, χρηματοδότησης. Οπότε αυτό που λέει η Κομισιόν είναι ότι εντάξει να υπάρχουν αυτοί η, αυτή η ατζέντα για την, για την ισότητα επί αλλά ε, στην πράξη τι γίνεται. Η Κομισιόν λοιπόν νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να το δει αυτό. Ε, το προσωπικό της Κομισιόν ε, βλέπουν, βλέπει φαντάζομαι την ε, αντίθεση και θα το πάρει σοβαρά υπόψη του. Αλλά όντως, πρέπει πολύ σοβαρά να δείτε το επίπεδο πόρων που χρειάζεται, ώστε έτσι να γίνει πράξη η ισότητα, να την προωθήσουμε, να μπορέσουμε να πιέσουμε στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της ισότητας πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο χρηματοδότηση για να μπορούν αυτοί οι αφορέ να λειτουργήσουν. Γιατί αλλιώ δεν έχει νόημα. Νομίζω λοιπόν, ε, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την ε, Ιρλανδική κυβέρνηση να έρθει εδώ ενώπιον τη Επιτροπή μα και να μα δώσει απαντήσει για τι πράξει τη. Γιατί νομίζω ότι πραγματικά ε, είναι εξόφθαλμο το πράγμα αυτό που πρέπει να μας απαντήσει. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις, μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αρχή ισότητας έχει κατά κάποιο τρόπο τιμωρηθεί, όχι επειδή ήταν αδύναμη, αλλά επειδή ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική και δραστήρια. Αυτή είναι η άποψή μου αφού άκουσα τα σχόλια της αναφέρουσας αλλά και από την Κομισιόν. Οπότε, αυτό δεν έχει συμβεί σε καμιά άλλη χώρα, στη δική μου Ρουμανία, όπου οι αρχές καθημερινά παραβιάζουν δικαιώματα και κανόνες, αλλά στην Ιρλανδία και κατά την άποψή μου αυτό είναι απαράδεκτο. Σε μια φάση οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης οι διακρίσεις και η, και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνεται καθημερινή πραγματικότητα. Τραγωδία. Ο κόσμος της Ευρώπης χρειάζεται μια αρχή, μια ανεξάρτητη αξιόπιστη ε, αρχή για να υπερασπιστεί και να προστατεύσει και να προωθήσει τα δικαιώματά του. Αλλά δεν χρειάζεται περικοπές στους σπόρους και στο ανθρώπινο δυναμικό τέτοιων αρχών ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των λαών της Ευρώπης, εάν δούμε τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε κάθε χώρα στην Ευρώπη. Οι ηλικιωμένοι υπόκειται σε διακρίσεις. Οι νέοι επίσης. Κατά κάποιο τρόπο και οι μειονότητες το ίδιο Ποιος, πού είναι ο δικαστής, πού είναι ο κριτής που θα προστατεύσει και θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά τους, ε, όχι μόνο στην Ιρλανδία αλλά και σε άλλο σωρό άλλα μέρη. Παρακαλώ λοιπόν να μην ανοιχτεί αυτή ε, η αναφορά και να μην είμαστε επίκης. Εντάξει, είναι, υπάρχει οικονομική κρίση και άρα πρέπει να δεχόμαστε ότι να είναι περικοπές και να συμμαζέψουμε τα οικονομικά. Τρία εκατομμύρια ευρώ είναι τόσο πολλά για τον ελλαδικό προπολογισμό ώστε δηλαδή αυτή η εν λόγω αρχή να πάψει τη λειτουργία της, να αναστείλει τελείω τη λειτουργία της. Εγώ ζητώ λοιπόν να στείλουμε μια επιστολή στην Ιρλανδική κυβέρνηση από εδώ από την Επιτροπή μας και να ζητήσω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι, ε, να, ε, να είναι άγρυπνη, να φροντίσει και να εξετάσει σοβαρά πώς λειτουργούν οι παρόμοιες αρχές στην Ευρώπη, διότι εδώ μιλάμε για τα ευρωπαϊκά δικαιώματα δικαιώματα που πρέπει να προστατεύονται από αρχές που έχουν δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είναι δική μας υποχρέωση και ευθύνη να φροντίσουμε ώστε να λειτουργούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Μποστινάρο. Πρόταση λοιπόν που νομίζω υποστηρίζουν όλοι είναι να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά και ταυτόχρονα να στείλουμε στείλουμε μία επιστολή στις Ιρλανδικές Αρχές για να λάβουν υπόψη αυτήν την περικοπή. Μάλλον να ζητήσουμε και να ρωτήσουμε πώς θεωρούν ότι θα λειτουργήσει αυτή η αρχή και πώς θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από, από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με αυτές τις περικοπές. Και θα περιμένουμε και την, ε, τα αποτελέσματα των τελευταίων ε, των τελευταίων πληροφοριών που θα μας δώσει η Κομισιόν. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο που είναι οι δύο ε, αναφορές στο σημείο 12 είναι η 997 2007 και η 15-18-2008. Είναι παρούσες οι, δύο, οι παρόντες οι δύο αναφέροντες. Είναι εδώ η Ειρήνα Ματέβα. Ναι, είμαι εδώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με κάλεστε σήμερα εδώ, σε αυτή τη συνεδρία της Επιτροπής αναφορών. Έχουν περάσει τρία, πάνω από τρία χρόνια από τότε που ε, η Βουλγαρία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από δυόμιση χρόνια που υπέγραψε την, ε, ε, το ψήφισμα για την προστασία των πτηνών. Το αίτημα, το, η αναφορά 997 για το, από το 2007 μιλά για την ανεπαρκή προστασία των, του δικτύου Natura 2000. Και το, η αναφορά 15-18 από το 2008 μιλάει για την ανεπαρκή προστασία των, ε, ε των ζωνών ε, της Natura 2000 ε, κοντά και στην προστασία των φτηνών κοντά στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουν υποβληθεί πολλά αιτήματα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ίδιο θέμα. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διάφορες διαδικασίες και έχουμε στείλει και έχει στείλει αρκετέ κοινοποίησει ε, στι βουλγαρικέ αρχέ. Παρ' όλα αυτά, οι δράσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα δεν ήταν αποτελεσματικέ ώστε να ε, αναγκάσει τη βουλγαρική κυβέρνηση να ε, συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία του Natura 2000. Να τονίσω επίση ότι θα έπρεπε να έχει, η, το, η περιοχή για την οποία σα μιλώ θα έπρεπε να έχει μπει στο Natura 2000 και ακόμη δεν έχει γίνει αυτό από το Δεκέμβριο του 2009 μόνο δύο καινούριε ε, περιοχές θεωρούνται ε, Natura 2000 και μόνο 90 από τις 114 επίσης θεωρούνται Natura 2000 και δεν, έχουν ληφθεί καμία, δεν έχει ληφθεί καμία δράση από, την, ε, από τις βουλγαρικές αρχές για να μπουν αυτές οι έξι περιοχές που βλέπετε στην οθόνη σας στο Natura 2000. δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια. Η ζημιά που έχει γίνει στη Βουλγαρία και στην φυσική της κληρονομιά δεν έχει διορθωθεί. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα των οικοσυστημάτων που καταστρέφονται σε μια περιοχή που προτείνεται αλλά δεν έχει καθοριστεί ως, καταχωρηθεί ως προστατευόμενη περιοχή. Εκεί υπάρχουν ε, σχέδια για να γίνει η μεγάλη ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη ε, Σημεία δηλαδή όπου, που πραγματικά μειώνουν, ε, συμπτύσσουν πάρα πολύ τις, ε, τα οικοσυστήματα. Έχει γίνει ζημιά που δεν αναστρέφεται σε, άλλο ένα, σε άλλη μια περιοχή, στον Πελή Τίσκαλη, ε, στην ε, ζημιά στο οικοσύστημα και από το 2006 η περιοχή αυτή βλέπετε πως ήταν εδώ στην οθόνη και τώρα ο... το οικοσύστημα έχει καταστραφεί παντελώς. Η, τα σημεία αυτά για τα οποία σας μιλώ είναι πολύ σημαντικά στη φορά τη ζωή των πτηνών και πάλι θα αναφερθώ στην καλή άκρα. Δύο χρόνια μετά την δημιουργία αυτού του αεολικού πάρκου δεν μπορεί να ε, επανασυγκροτηθεί ο οικότοπος και έχει γίνει απλώς μια έρημος και δεν μπορεί να γίνει καμία ε, δεν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση πια. Επίσης, ε, χτίζεται μια καινούργια φάρμα, ένα καινούργιο ολικό πάρκο με γερμανική εταιρεία η οποία επενδύει στο έργο. Και αυτή, αυτό το ολικό πάρκο η κυβέρνηση προσπάθησε να το σταματήσει αλλά το αποτέλεσμα της ε, απόφασης δεν ήταν καταληκτικό. Επίσης, τον Γενάρη του 2010 ξεκίνησε να λειτουργεί ένα μεγάλο ορικό πάρκο σε μια περιοχή η οποία προτείνεται αλλά δεν έχει καταχωρηθεί ως περιοχή Natura 2000 η οποία επίσης παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η βουλγαρική κοινότητα προστασία των πτηνών είναι πολύ ικανοποιημένη που η Κομισιόν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάση. Αλλά η βουλγαρική κυβέρνηση δεν δείχνει καμία διάθεση να αλλάξει την προσέγγιση τη παρά τι δράσει που έχουν γίνει μέχρι στιγμή. Έγιναν κάποιε προσπάθειε να ενισχυθεί η διαδικασία τη έγκριση των νεολικών πάρκων ώστε κάθε ολικό πάρκο να υπόκειται σε περιβαλλοντική αξιολόγηση επιπτώσεων. Η κυβέρνηση προσπάθησε να, κάνει, να επιβάλλει μορατόριουμ στις ε, κατασκευές ολικών ε, πάρκων, αλλά απέτυχαν όλες αυτές οι προσπάθειες. Η πρόσφατη αλλαγή στην κυβέρνηση δεν ε, άλλαξε κάτι σε ό,τι αφορά τις περιοχές που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πρέπει να προστατεύονται. Υπάρχει και η νομοθεσία για την προστασία των απτηνών, υπάρχει και σχετική οδηγία η οποία έχει θέσει και κάποιους ευρωπαϊκούς στόχους που πρέπει να ε, πραγματοποιηθούν. δεν μπορούν τα κρατημέλη λοιπόν να, την, να διαφορούν για την οδηγία. Είναι λοιπόν ώρα η Κομισιόν να αναλάβει δράση, να στείλει δεν έχει νόημα να στέλνει άλλε προειδοποίησει ε, ή να συμφωνεί με τι ε, υποσχέσει που τη δίνει η βουλγαρική κυβέρνηση. Νομίζω ότι θα πρέπει η ε, Κομισιόν να, επιβάλλει, να δώσει γνωμοδότηση εναντίον τη Βουλγαρία για, για τη μη συμπερίληψη κάποιων περιοχών στο Natura 2000. Να ξεκινήσει μια διαδικασία στο δικαστήριο, έτσι ώστε να δούμε πώ έχει γίνει η καταστροφή στην περιοχή αυτή, την Καλιάκρα και να γίνει και, συνα... και ε, συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων. Η καταστροφή συνεχίζεται σε όλες τις περιοχές που θα έπρεπε να είναι στο Natura 2000 στη Βουλγαρία και δεν είναι. Οι περιοχές αυτές, βέβαια για τις περιοχές αυτές μάλλον η Κομισιόν μπορεί να μην έχει δυνατότητα να λάβει δράση και θα ήθελα να σας ζητήσω εδώ στην Επιτροπή Αναφορών ε, να πιέσετε και σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να σας, να σας αναφέρω ποια είναι τα προβλήματα στη Βουλγαρία και πραγματικά θα ήθελα να παρακολουθήσετε το τι θα γίνει με την ε, αναφορά αυτή. Επίση, ε, θα πρέπει ίσω να έρθουμε και σε επαφή με τον ε, Επίτροπο περιβάλλοντο για να δούμε κατά πόσο μπορεί να αναλυθεί μια δράση περιβαλλοντική στη Βουλγαρία και να τονίσουμε την ανάγκη για επαρκείς πόρου οι οποίοι θα πρέπει να επενδυθούν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη νομοθεσία. Ίσως και να πρέπει και μια αποστολή να επισκεφθεί τη Βουλγαρία. Εμεί ευχαρίστω να σα ε, φιλοξενήσουμε ώστε να μπορέσετε κι εσείς να δείτε πώς έχει η κατάσταση επιτόπου. Επίσης ε, να καλέσουμε τον ε, Βουλγαρό Υπουργό Περιβάλλοντος να έρθει εδώ, να τον καλέσετε αν θέλετε, να έρθει εδώ στην Επιτροπή Αναφορών, ώστε να του δώσετε ποια είναι η, να, του, να, δώσετε και να δείτε ποια είναι η προσέγγιση της α, ε, α, βουλγαρικής κυβέρνησης ό,τι αφορά την εφαρμογή της α, περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως θα γνωρίζετε, οι αναφορές αυτές έχουν συζητηθεί και άλλη φορά εδώ. Οπότε θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω κάπως, ιδίως σε σχέση με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που ακούσαμε μόλις τώρα από την αναφέρουσα. Όπως υπογράμισε, οι δύο αναφορές είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στρατηγικής σημασίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τους ε, οικοτόπους στη Βουλγαρία. Αναφέρεται σε διάφορες διαδικασίες επιπαραβάση που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα προσπαθήσω εδώ να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές κλειδί που περιλαμβάνονται στις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχετικές αναφορές. Αν δούμε το θέμα του ορισμού των ε, χώρων. Πρώτα απ' όλα ορίζονται βάσει της οδηγίας ΠΑΤΣ και στη συνέχεια έχουμε την αναγνώριση των χώρων βάσει της οδηγίας Habitat για τους οικοτόπους. Βάσει της πρώτης οδηγίας η Βουλγαρία έχει ορίσει όλες τις περιοχές που εντοπίστηκαν από τη Βουλγαρία. Όμως υπάρχει εδώ ένα ζήτημα για μερικές περιπτώσεις. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανταλλαγή απόψεων με τις αρχές της Βουλγαρίας προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο η οριοθέτηση των περιοχών προστασίας έχει γίνει ορθά και πλήρως. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή, γιατί πρέπει να ελέγξουμε πολλά είδη, πολλές αναφορές. Πάντως μετά από τις συζητήσεις που είχαμε και λαμβάνοντα υπόψη πληροφορίες που μας έδωσε και η αναφέρουσα, θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε παρετέρω μέσα στους επόμενους μήνες. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί δεν μπορώ να προκαταλάβω ποια ακριβώς θα είναι η θέση που θα υιοθετήσουν ε, οι επίτροποι. Όμως δουλεύουμε πάνω σε αυτό και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και τους επόμενους μήνες. Έτσι ερχόμαστε τώρα στην ε, αναγνώριση των περιοχών βάσει της οδηγίας Habitat. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι όπως και παλιότερα διαπιστώνουμε ότι η Βουλγαρία έχει παρουσιάσει ένα μεγάλο ποσοστό της επικράτειά της να συμπεριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσοστό. Και αυτή είναι μια παρατήρηση που έχει τη σημασία της νομίζω. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι έχει τελειώσει η δουλειά. Εδώ ο συνάδελφος Φώτης Παπούλιας θα σας πει σε λίγο δύο λόγια για το που βρισκόμαστε με τη διαδικασία που διασφαλίζει ότι όλοι οι κότοποι και όλα τα είδη καλύπτονται πλήρως. Περνώ τώρα στην πτυχή που έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι όλες αυτές οι περιοχές προστατεύονται ικανοποιητικά. Η αναφέρουσα πολύ σωστά αναφέρθηκε στις διαδικασίες επί που έχουν ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια διαδικασία επί παραβάση όσον αφορά την περιοχή Καλιάκρα που ανέφερε μόλις τώρα η αναφέρουσα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα στρατηγικής σημασίας για ένα γενικότερο πρόβλημα που έχει να κάνει με μη αξιολόγηση των επιπτώσεων όσον αφορά τις εξελίξεις στις περιοχές αυτές. Και γι' αυτό και έχουμε στείλει επιπλέον επιστολή στη Βουλγαρία το Μάρτιο. Πρέπει να ελέγξουμε τα στοιχεία. Χρειαζόμαστε επιπλέον επιστημονικά δεδομένα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις διάφορες περιπτώσεις όπως αυτή και άλλες περιπτώσεις ε, πήγανε στο δικαστήριο. Κάναμε εμείς δηλαδή προσφυγές και προσπαθούμε να πείσουμε το δικαστήριο ότι τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αρκετά για να οδηγήσουν ε, σε καταδίκη του κράτους μέλους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε να είναι πάντα αρκετά, ώστε να μπορεί να πιστεί το δικαστήριο. Πάντως συνεχίζουμε να εξετάζουμε τις περιπτώσεις αυτές και εφόσον χρειάζεται το Σώμα των Επιτρόπων θα δώσει συνέχεια με διαδικασίες τους επόμενους μήνες. Πέρα τώρα από τις διαδικασίες επί παραβάση, είχαμε και συζητήσεις με τις βουλγαρικές αρχές, προσπαθώντας να πείσουμε τη Βουλγαρία για το πόσο μεγάλη σημασία έχει η βελτίωση των διαδικασιών όσον αφορά την προστασία των χώρων αυτών. Τον Μάρτιο λοιπόν οργανώσαμε ένα σεμινάριο στη Σόφια με αξιωματούχους της Βουλγαρίας για να εξηγήσουμε τους κανόνες που εφαρμόζονται στους χώρους, της περιοχές της Natura 2000 για να ευθυγραμμιστεί και η Βουλγαρία με τις δύο οδηγίε. Περιμένουμε λοιπόν ότι θα συνεχίσει η Επιτροπή να ασχολείται και θα σας ενημερώνουμε για την πρόοδο που επιτυχάνεται όσον αφορά τις αναφορές αυτές. Ο συνάδελφός μου Φώτης τώρα θα πάρει το λόγο για να σας πει πού βρισκόμαστε όσον αφορά την αναγνώριση των περιοχών βάσει της οδηγίας Habitat. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να προσθέσω μερικά στοιχεία για την αναγνώριση περιοχών υπό την οδηγία Habitat. Πρόκειται για τις λεγόμενες ε, σημαντικές ε, περιοχές. Πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε με ένα βιογεωγραφικό σεμινάριο για την περιοχή και παρά το σημαντικό ποσοστό της επικράτειας που είναι 30% υπήρχαν κάποια κενά που εντοπίστηκαν. Οι αρχές ανάλαβαν την υποχρέωση να καλύψουν τα κενά αυτά από τη μια και από την άλλη να αναλάβουν, να εκπονήσουν επιστημονικές μελέτες με έρευνες ώστε να διευκρινιστεί η κατάσταση. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2008 έχουν ήδη καλυφθεί κάποια μικρά βέβαια κενά αλλά για τα πιο μεγάλα που χρειάζεται ακόμα δουλειά, για 36 ήδη για παράδειγμα, χρειάζονται ευρύτερες έρευνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως έχει συνεχώς επαφές με τις βουλγαρικές αρχές και συμφώνησε να δώσει περισσότερο χρόνο στη Βουλγαρία ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει ε, σωστά τις έρευνες και τα κενά που υπήρχαν μέχρι τώρα. Το συμφωνήσαμε λοιπόν αυτό και πάμε έτσι μέχρι το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο του 2010. Μετά από τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επαναξιολογήσει τον ορισμό των περιοχών αυτών, κατά πόσο είναι σωστός ή όχι. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Πριν δώσω το λόγο στην αναφέρουσα και πάλι. Θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Παστινάρουσε το λόγο και η κυρία Χόκαν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας τα πω αγγλικά καλύτερα. Να δούμε τα στοιχεία, όχι μόνο τις εικόνες, αλλά και τις στατιστικές. Το περιεχόμενο της αναφοράς επιβεβαιώνει, δυστυχώς, τα συμπεράσματα της έκθεσής μας για τη βιοπικιλότητα. Αυτό είναι γεγονός. Δεύτερον, δεν είναι μόνο μια επιβεβαίωση, αλλά και μια επιδεινούμενη κατάσταση που, λέει, που μας δείχνει ότι όταν οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένουν υπερβολικά πριν να προβούν σε δράση, όχι μόνο είναι πολύ αργά, αλλά πολύ συχνά είναι ανα... Ε, δεν είναι αναστρέψιμη πια η κατάσταση. Και βλέποντας τις εικόνες από την καλλιάκρα με εκείνο το αιωλικό πάρκο και τη σχετική υποδομή που έχει απεριμωθεί η περιοχή, τι περισσότερα στοιχεία χρειαζόμαστε πριν να δράσουμε. Τρία. Ορισμένες φορές οι εθνικές κυβερνήσεις είναι υπερβολικά αδύναμες όταν ε, αγωνίζονται κατά μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, κατά μεγάλων πολυεθνικών φορέων, όταν αγωνίζονται κατά πολυεθνικών εταιριών. Γιατί εδώ πρόκειται για χρήματα και κέρδη για τα κέρδη μεγάλα. Και η κυβέρνηση είναι υπό τεράστια πίεση από τη μια πλευρά. Έχουν την οικονομική κοινότητα, δηλαδή τους επενδυτές, και από την άλλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητά από το Βουκουρέστι, τη Σόφια ή οποιαδήποτε άλλη πρωτεύουσα και λέει παρακαλώ κάντε κάτι αλλά πριν ενεργήσετε πριν μάλλον ενεργήσουμε είναι πια πολύ αργά. Και μια τελική μου έκκληση προς την Επιτροπή. Χρειάζεται μέσα στο νέο πλαίσιο όταν η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα υιοθετήσει την έκθεσή της για την βιοπικιλότητα, χρειάζονται χρονικά όρια για τις δράσεις των εθνικών κυβερνήσεων και για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί διαφορετικά θα παρακολουθήσουμε παθητικά πώς καταστρέφουμε τη φύση πως πώς βυθίζουμε την, κατα, την βιοπικιλότητα της Ευρώπης, πώς καταστρέφουμε τη βιοπικιλότητα. Δεν χρειάζονται άλλες μαρτυρίες. Έχουμε αρκετές αποδείξεις για να ενεργήσουμε. Νομίζω πως η βουλγαρική περίπτωση και όχι μόνο η βουλγαρική και πολλές άλλες χρειάζονται χρονικά όρια για δράση και όχι μόνο για εξηγήσει που δεν είναι καθόλου αποτελεσματικές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρο. Κυρία Όκ. Υποστηρίζω απόλυτα αυτά που είπε ο συνάδελφος. Είναι όντως πολύ σημαντικό να Ξέρουμε ότι η Κομισιόν είναι πολύ αδύναμη με αυτή την οδηγία και απλώς ακολουθεί κάποιες μεγάλες δυνάμεις. Αν δεν απαντήσουμε τώρα θα υπονομεύσουμε τη δουλειά μας, τη δουλειά που έχουμε κάνει για να υποστηρίξουμε, να προστατεύσουμε το Natura 2000. Οπότε υποστηρίζω αυτά που λέτε και μήπως θα έπρεπε να κάνουμε όντω μια αποστολή στη Βουλγαρία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε και στην παράκτεια περιοχή και στην Μαύρη Θάλασσα. Εγώ πριν από δύο χρόνια πήγα και πραγματικά είναι απερίγραπτο το πόσα πράγματα δεν λαμβάνουν σοβαρά οι βουλγαρικές αρχές. Και απ' την άλλη, ο πληθυσμός γνώριζε πολύ καλά. Υπήρχε μεγάλη ευαισθητοποίηση. Θέλουν να κάνουμε κάτι εμείς. Δεν είναι ε, ένας παραμελημένος πληθυσμός. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Ίσως λοιπόν έπρεπε να στείλουμε μια αποστολή στη Βουλγαρία για να δούμε επιτόπου το τι γίνεται. Eh, Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλος το λόγο, δεν ξέρω. Ποιος άλλος. Α, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτό που, είπε, που είπαν οι συνάδελφοι, ο διάλογο μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών θα πρέπει να ξεκινά νωρί. Και σε ό,τι αφορά το Natura 2000 και το Habitat, ε, την προστασία των πτηνών, την οδηγία πλαίσιο. Ε, πρέπει να ξεκινούμε δηλαδή με κάτι θετικό. Είναι προς ε, το συμφέρον του κράτους μέλου να ξεκινάει νωρί ο, ο, διάλογος για να μην αρχίζουν τώρα και μπαίνουν καθυστερήσει μέσα και τραβάει το πράγμα. Ξεκινούμε λοιπόν εμείς την πρώτη φάση, ξεκινούμε τη δουλειά και αν όντως υπάρχουν στοιχεία ότι α, υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας κτλ. τότε μπορούμε να δράσουμε. Οπότε δεν είναι μόνο προς όφελος της τάξης, είναι προς όφελος της Κομισιόν, είναι προ όφελο του Κοινοβουλίου, αλλά κυρίω είναι προ όφελο του κράτου μέλου. Νωρί να ξεκινούμε το διάλογο, έτσι ώστε να μην τραβάνε οι διαδικασίε αυτέ ε, επί Γιατί υπάρχουν και πολλά θέματα που άπτονται ε, δύο κρατών μελών, γιατί οι περιοχέ που συζητούμε είναι στα σύνορα. Οπότε καταρχήν να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα πράγματα γίνονται τυπικά και αν δούμε ότι όντως υπάρχουν παραβιάσεις, παρανομίες και όταν, τις παρουσια... όταν δούμε τις παρανομίες τότε να πρέπει να δράσουμε ίσως τότε όμως δεν είναι πολύ αργά γιατί αυτή είναι και η συνήθις πρακτική τώρα ίσως λοιπόν να πρέπει νωρίς να ξεκινούμε και από τις πρώτες κιόλας συνδείξεις να δρούμε Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την αναφέρουσα που μας παρουσίασε τόσο ξεκάθαρα ποιο είναι το πρόβλημα στη Βουλγαρία. Στηρίζω την ιδέα της για το ότι πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο στις αναλύσεις μας και κάτι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να αναφερθώ σε δύο πράγματα στο διάλογο. Ο διάλογος πριν από το 2007 δεν υπήρχε. Οι προθεσμίες μίκρυναν για τις επαφές βουλγαρικής κυβέρνησης με την Κομισιόν. Η νέα κυβέρνηση λοιπόν έχει ήδη εκφράσει τη βούλησή της να διορθώσει το πρόβλημα που υπενθυμίζω έχουμε ημερομηνίες από το 2008 και 2009. Έπειτα, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ορισμένα προβλήματα, για ορισμένα θέματα πρέπει να περιμένουμε το τέλος της χρονιάς αυτής. Οπότε, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να διονυστεί η υπόθεση. Φυσικά και πρέπει κάτι να κάνουμε, πρέπει να δράσουμε, αλλά υπογραμμίζω ότι από τότε που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση το 2009, ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεκαταστάθη, επιταχύνθηκε, καθορίστηκαν πολύ συγκεκριμένες προθεσμίες, όπως ε, εκείνη του Οκτωβρίου του 2010. Η νέα λοιπόν κυβέρνηση έχει δηλώσει βούληση. Και το επενθυμίζω, μερικές φορές είναι δύσκολο να βρούμε μια λύση σε προβλήματα οικονομικών συμφερόντων και ευχαριστώ τον συνάδελφο που το έθεσε. Βλέπετε ορισμένε άδειε οικοδόμηση δόθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πώ να τι αποσύρουμε τώρα με νόμιμο τρόπο. Καταλαβαίνετε και αυτοί έχουν τα επιχειρήματά του. Οπότε πρόκειται για καταστάσει πολύ λεπτέ και δύσκολε. Όμω, ω εκπρόσωπος και εγώ της κυβέρνησης που έχει την εξουσία σήμερα στη Βουλγαρία, σας επιβεβαιώνω ότι είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και έτοιμοι από κοινού να βρούμε λύσεις. Ευχαριστώ πολύ πάνω από όλα αυτούς τους τόσο ενεργούς ε, βούλγαρους πολίτες που δηλώνουν τη δικιά τους βούληση να προστατεύσουν το φυσικό μας περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση η αναφέρουσα να πάρει και πάλι το λόγο εφόσον θέλετε κάτι να προσθέσετε. Έχετε κάτι να πείτε. for your comments. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Το μόνο πράγμα που θέλω να προσθέσω είναι ότι η κατάσταση επήγει Χρειάζονται από κοινού δράσεις από την βουλγαρική κυβέρνηση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά που είδατε έγιναν ανάμεσα στην πρώτη μας αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών εδώ και τώρα. Κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα χειροτερεύουν οι δράσεις της νέας κυβέρνησης έχουν να κάνουν πιο πολύ με το μέλλον. Δεν ε, διορθώνουν το σημερινό πρόβλημα. Και αν δεν κάνει κάτι περισσότερο για το σημερινό πρόβλημα θα καταστραφεί το περιβάλλον. Πράγματι είναι λεπτό και δύσκολο να λυθούν τέτοια προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, αλλά πρέπει να αναλυφθούν δράσεις και να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα για να καταλήξουμε σε μια καλή λύση όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι όλοι όσοι πήραν το λόγο έδειξαν ότι καλό θα ήταν να μείνει ανοιχτή η αναφορά και ο γραμματέα που ξέρει μερικέ φορέ περισσότερο και από εμά. Γιατί εμεί οι βουλευτέ βλέπετε ερχόμαστε εδώ χωρί γραβάτα ενώ βλέπετε πόσο σοβαρό είναι εδώ ο γραμματέα με τη γραβάτα του. Μου λέει λοιπόν ότι ίσω θα έπρεπε να το δει το θέμα αυτό και η Επιτροπή Περιβάλλοντος για να τη μελετήσει την αναφορά αυτή και η Επιτροπή περιβάλλοντο και να βοηθήσει και εκείνη την αναφέρουσα, όπως έλεγε και η κυρία Μιλαντσέβα, την οποία και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την αναφέρουσα που ήρθε από τη Βουλγαρία, μας μετέφερε τις ανησυχίες της και ελπίζουμε να λυθεί. Και όχι μόνο από εμά, αλλά εφόσον συμφωνείτε και εσείς, οι ευρωβουλευτές εδώ, να ζητήσουμε και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος να παρέμβει. Καλώ. Ωραία. Το σημειώνουμε. Και περνάμε τώρα στην οδηγία 13. Σημείο 13, λοιπόν. Τα έχω δώσει τα ιταλικά, βλέπετε. Είναι η 7, Είναι 7, 2009 του Πάτρικ Κίνεσλι εξ ονόματος ε, της συμμαχίας White Horse σχετικά σχετικά με την εικαζόμενη παράληψη των Βρετανικών αρχών να συμμορφωθούν με την κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη παρακαμπτήρια εδώ του και άλλα οδικά προγράμματα. Σχέδια. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κίνινες, λοιπόν είναι παρόν. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως εισαγωγή έχετε μια εικόνα του λευκού ύπου στο Westbury ως κομμάτι των πληροφοριών που θα σας δώσουμε μέσω των διαφανειών που έχουμε. Ευχαριστώ την Επιτροπή Αναφορών που δέχτηκε την αναφορά μας και την Εκτελεστική Επιτροπή που συνέταξε μια τόσο επικοδομητική και βοηθητική επιστολή προς την Επιτροπή σας. Έχω συντάξει αυτήν την δήλωση Ελπίζοντα πως θα βοηθήσει την Επιτροπή στις διαβουλεύσει τη και ζητώ συγγνώμη που είναι τόσο μακρά η δήλωση αυτή. Θα προσπαθήσω, στην γραπτή της μορφή, θα προσπαθήσω να αναφέρω σύντομα τα κεντρικότερα σημεία γιατί ξέρω πως ήδη έχετε καθυστερήσει. Αλλά και επίσης επειδή θέλουμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Επιτροπή. και ίσω να ακούσουμε για κάποια παρέμβαση ίσως και κίνηση διαδικασία επί παραβάση από πλευρά τη Κομισιόν. Θα ήθελα να σα παρουσιάσω τη συνάδελφο Jenny Ράγκετ που προετοίμασε το ε, οπτικό υλικό της είναι και εκείνη στη Διοικητική Επιτροπή της ε, συμμαχία για του Λευκού Ήπου που σχηματίσαμε πριν από δύο χρόνια περίπου για να αγωνιστούμε κατά της παρακαμπτηρίου του Westbury. Επίσης ήταν ε, μέλος ε, της συνέλευσης της νοτιοανατολικής περιφέρειας και έχει γίνει και η τελευταία έκθεση μάλλον ε, δοκιμή περιβαλλοντικών επιπτώσεων και από ό,τι φαίνεται τα κρατημέλη το κράτος μέλος δεν έχει φτιάξει ένα σύστημα ώστε να εξασφαλίσει συμμόρφωση προς την οδηγία περί κοτόπων. Αν η απλούστερη ερώτηση είναι κατά πόσο μία υπηρεσία, κάποιος οργανισμός ε, υποχρηματοδοτούμενος μπορεί να πει ναι ή όχι, τότε εντάξει, αλλά το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό. Υποβάλαμε αυτή την ε, αναφορά πριν από ένα χρόνο όταν ε, θεωρήσαμε πως αυτή, αυτό το σχέδιο θα προχωρούσε αναπόφευκτα γιατί το επιθυμούσαν όλα όλοι οι φορείς, οι αρμόδιοι φορείς του κράτους μας και δεν υπήρχε καμία αντίσταση από πλευρά της υπηρεσίας φύση, φύση και Αγγλία και ήταν σίγουρο ότι αυτό παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας περί για την προστασία των ειδών αλλά και ε, την προστασία των τοποθεσιών του Natura 2000. Αυτό εδώ είναι το τοπίο που μπορείτε να δείτε. Ασβεστούχοι λόφοι είναι, που μπορείτε να δείτε είναι αυτοί οι οποίοι πρόκειται να αλλοιωθούν. Το ασβέστιο έχει εξοριχθεί μέσω εξόριξης για να δείξουμε τον λόφο του λευκού ύπου. Πρόκειται για τεράστιες όγκους ε, ασβεστίου που θα εξοριχθούν και πράγμα το οποίο θα λιώσει τελείως αυτό το, την κληρονομιά που μπορείτε να δείτε στην οθόνη. Η επιπτώση στο περιβάλλον ε, ήταν εμφανής εξ αρχής. Η άποψή μας είναι πως είναι μια δοκιμή αυτή. Για να, για, που λέει ότι αν μπορείς να φτιάξεις ένα δρόμο εδώ, μπορείς να κατασκευάσεις και δρόμο οπουδήποτε αλλού. Και είμαστε αποφασισμένοι να το σταματήσουμε. Μπορείτε να δείτε από τις εικόνες. Καταρχήν, πως το τοπίο και κληρονομιά του, του, της τοποθεσίας White Horse που είναι από την εποχή του Σιδήρου τα πρώτα σημεία ζωής καθώς και όλες τις περιοχές της τοποθεσίας ε, γύρω αναγνωρίστηκε από το 1951 μετά από τον πόλεμο όταν ε, η Εθνική Επιτροπή Δρυμών σύστησε να αποτελέσει αυτός ο χώρος εθνικό δρυμό ή χώρο εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς. Δυστυχώς το τοπίο δεν προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό έχει να κάνει με το ότι η ιδιοκτησία είναι του Υπουργείου ε, Αμήνης και αυτό το Υπουργείο έχει αντισταθεί στον χαρακτηρισμό της περιοχής ως ε, προστατευόμενης. Επίσης υπάρχουν ε, υδάτινοι πόροι που είναι προστατευόμενοι σε αυτή την κοιλάδα και, φυσικά, και κανονικά κάτι τέτοιο θα σταματούσε τα σχέδια γιατί αυτή η υδάτινη πόρη είναι πολύ σημαντική και για την άγρια ζωή και όχι μόνο ως ε, λεκάνη παροχής ύδατος στον πληθυσμό. Η σημασία της βιοπικιλότητας επίσης θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρη από την αρχή, όμως η κοιλάδα του Σέλσμπουρη δεν υπήρχε, που είναι επίσης ε, προστατευόμενη, δεν ενέπιπτε μέσα στις ε, περιοχές, ε, στις περιοχές προστασίας. Και το Συμβούλιο Natural England, που είναι η αρμόδια υπηρεσία, δεν αποφάσισε να συμπεριληφθεί εκεί. Ούτε θεωρήθηκε ειδική περιοχή προστασίας και συντήρησης. Συγγνώμη, πρέπει να πιω λίγο νερό. Ε, okay. Um. Ε, Πιστεύουμε πως εξ αρχής θα έπρεπε να έχει γίνει μια σωστή αξιολόγηση λόγω των δύο ειδικών περιοχών προστασίας και ιδιαίτερα το Μπάθ και το Bradford των Avon που είναι προστατευόμενες περιοχές. Όμως αυτή η αξιολόγηση δεν έγινε και τελικά παρενέβη το Ευρωπαϊ... Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προστασίας Νυχτερίδων. Αρχικά η αρμόδια υπηρεσία ε, έφερε αντιρρήσεις στο πρόγραμμα και προσέφερε κάποιες προτάσεις άβλησης του τον αντικτύπου ε, ώστε αυτός να φτάσει σε ένα επίπεδο ενός μικρού ε, αντικτύπου, εν πάση περιπτώσει. Ο χάρτης δείχνει τι ήταν γνωστό από το 2003 και δημοσιεύθηκε το 2004. Ένας μεγάλος αριθμός ε, ειδών νυχτερίδων που συμπεριλαμβάνει και τρία είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2 της οδηγίας Ε, που είναι προστατευόμενα ήδη δηλαδή. Γνωρίζω το χρόνο, ναι, έχω πολύ κείμενο, πολύ κείμενο εδώ και προσπαθώ να το συντομεύσω, αλλά μάλλον δεν τα πάω και πολύ καλά. Πόσο χρόνο έχουμε? Sorry. Um... so I have problems with coordinating this presentation. Ναι, έχω πρόβλημα να συντονιστώ με αυτή την παρουσίαση. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε ότι κανονικά το σχέδιο αυτό θα είχε, πρέπει να έχει λάβει υπόψη τη σημασία της άγριας ζωής στην περιοχή και ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν έχουμε καταφέρει να το σταματήσουμε γιατί πολύ λίγοι δρόμοι σταματούν. Τον Ιούλιο του 2009 μάθαμε ότι είχαμε καταφέρει κάτι άνευ προηγουμένου. Σταμάτησε το πρόγραμμα, σταμάτησε το σχέδιο γιατί ο επιθεωρητής στην δημόσια έρευνα είπε ότι δεν μπορούσε να σταθεί αυτό εδώ το σχέδιο γιατί δεν δικαιολογούσε τη σημαντική ζημιά που θα έκανε, θα επέφερε στον τοπικό στην, λόγο τοποθεσία. Η κυβέρνηση συμφώνησε, αλλά παρά τις αποδείξεις από επιφανείς οικολόγους που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, τελικά ούτε ο επιθεωρητής ούτε η κυβέρνηση αμφισβήτησαν την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι ο αντίκτυπος δηλαδή στην άγρια ζωή θα ήταν παράδειγμα. Καταφέραμε το στόχο μας να υπερασπιστούμε ε, έναν χώρο σπάνιας ομορφιάς και ηρεμίας, αλλά η οδηγία των οικοτόπων δεν έπαιξε ρόλο στην ε, διάσωση της άγριας ζωής ε, που ε, που υπάρχει σε αυτό τον σπάνιο οικότοπο. Ολόκληρη η οδηγία, μάλλον το παραθυράκι στην οδηγία περί οικοτόπων παραμένει ανοιχτό. Η ευρωπαϊκή άγρια ζωή είναι το ίδιο ευάλωτη όσο ήταν ανέκαθεν. Και από την εμπειρία μας στο Westbury, και στην νότιο-ανατολική, νοτιο μας περιφέρεια η, απλά είναι μία ακόμη απόδειξη της ευρείας αποτυχίας του Ηνωμένου Βασιλείου να ε, συμμορφωθεί προς την οδηγία περί οικοτόπων. Και από τότε που ελήφθη η απόφαση δεν έχουμε καταφέρει να να έχουμε περισσότερη προστασία. Καμιά ενθάρρυνση δεν μας έχει προέλθει από την Natural England που είναι το σώμα που είναι αρμόδιο για την προστασία του τοπίου και την προστασία των, της άγριας ζωής στην Αγγλία. Το Συμβούλιο της Κομιτείας που ξεκίνησε το σχέδιο αυτό τώρα συντάσσει περαιτέρω σχέδια για ανάπτυξη σε ολόκληρο τον ε, διάδρομο που ήταν μέρος του και αυτή η παρακαμπτήρια εδώ. Βλέπετε το βαθμό αυτού του σχεδίου στον χάρτη. Προχωρά από, είναι ο κόκκινος διάδρομος από την M4, τον αυτοκινητόδρομο M4, μέχρι την Α36, την Εθνική Οδό Α36 δείχνει επέκταση με βάση οδικό δίκτυο σε ένα μεγάλο κομμάτι της εξοχής και μία από αυτές τις περιοχές είναι εξαιρετικά σημαντική διότι έχουμε ένα νέο κομμάτι τμήμα 12 χιλιόμετρων του δρόμου Α35 ε, που θα παρακάμψει το δυτικό Άστον. Δεν ξέρουμε τώρα αν το πρόγραμμα αυτό θα προχωρήσει λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης αλλά ανησυχία μας είναι ότι το Συμβούλιο της Κομιτείας προτείνει να χρηματοδοτηθεί μέσω μιας ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας για ε, στεγαστικά σχέδια και βιομηχανικά σχέδια που θα ξεπεράσει το δυτικό ε, όριο του οδικού δικτύου και μπορεί να είναι τελείως αντίθετο μάλλον απέναντι από τα δάση Πίκετ και Κλάγκερ μία, ε, έναν αρχαίο δασότοπο όπου βρίσκουν καταφύγιο τεράστιες ε, ε, ομάδες από διάφορα σπάνια είδη. Τώρα βλέπουμε μέσω, ξέρουμε μάλλον, μέσω εντοπισμού από το καλοκαίρι του 2008 ότι υπάρχει μεγάλη σύνδεση ανάμεσα στα νυχτερίδες του Westbury και της προστατευόμενες περιοχές. Ο καθηγητής Τζον Άλτριχαν συνόψισε τις ε, επιπτώσεις των νέων στοιχείων που έχουμε συλλέξει στο εξή συμπέρασμα ότι η μεγάλη αναλογία νυχτερίδων που πιάνονται έχουν, ένα συστενό έχουν μια, έχει μια στενή σχέση με τα μεγάλα προβλήματα που απορρέουν από την απόφαση του να μην γίνει μια κατάλληλη αξιολόγηση επιπτώσεων. Κανονικά ε, το ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε την εκπόνηση ε, μιας αξιολόγησης επιπτώσεων, αλλά η αρμόδια υπηρεσία έχει εκφράσει αντίρρηση προς την ε, στρατηγική ανάπτυξη του Συμβουλίου του Wiltshire και για πρώτη φορά είδαμε μια αναφορά στην οδηγία για τους οικοτόπους όσον αφορά την χωροταξία. Επί τη βάση του ότι εκεί είναι ε, ε, περιοχές εκείησης των νυχτερίδων. Ναι, συγγνώμη, τα λέω πολύ αργά, ε, Πολ. Yes. If, if you can see the screen, the uh, questions that uh, the process that Jenny has um, uh, put, put onto this slide. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε νομίζω ξεκάθαρα τις ε, προσδοκίες που έχουμε εδώ στον σχεδιασμό και στη χωροταξία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τελικά όμως είναι το βασικό ερώτημα αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως ε, για την ε, νοτιοδυτική Αγγλία ότι δηλαδή η, η υπηρεσία φυσική Αγγλία δεν έχει αντισταθεί Χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης εξ αρχής ενώ τα περισσότερα σχέδια προχωρούν στην κατασκευή και μετά ε, ή δεν γίνεται καθόλου η αξιολόγηση αντικτύπου και πιστεύουμε πως αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν κινδυνεύει μια προστατευόμενη περιοχή από έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο ή κάποια άλλο σχέδιο. Σας ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα τόσο πολύ ναι, το θέμα είναι ότι μπορεί να μην έχουμε χρόνο για να πάρουμε τις απαντήσεις. Αυτό είναι. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Κάσμαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ο αναφέρον προσπάθησε να μας κάνει μια πολύ, να μας δώσει μια πολύ γενική εικόνα της αναφοράς του για το ποια είναι τα βασικά στοιχεία, μας μίλησε για τις αρμόδιες βρετανικές αρχές, οι οποίες ε, δεν έδωσαν το πράσινο φως στην ε, παρακαμπτήριο του Westbury. Και ότι αυτό ανησυχούσε τον αναφέροντα. Επίσης ε, μίλησε για την άρνηση της έγκρισης για την κατασκευή των οδικών ε, των ε, δρόμων που θα περάσουν από την περιοχή εκεί. Και μας μίλησε και για τις σκέψεις που έγιναν σχετικά με την κατασκευή των δρόμων αυτών ε, και στα πλαίσια της συμμόρφωσης με την οδηγία για τους οικοτόπους. Εμείς έχουμε ζητήσει διευκρινήσει από τι βρετανικέ αρχέ. Ελπίζουμε να τι λάβουμε μέσα στου επόμενου δύο μήνε. Μόλι θα έχουμε απάντηση, θα έρθουμε και πάλι σε επαφή με την Επιτροπή σα για να σα ενημερώσουμε για το ποια είναι η θέση των Βρετανικών Αρχών και σε σχέση με τις ανησυχίες που εξέφρασε ο αναφέρον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο άλλος κύριος Κάσμαν τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περίεργο ένας Κάσμαν να ακολουθεί έναν άλλο Κάσμαν, αλλά βλέπετε συμβαίνουν και αυτά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε εγώ θα πω απλώ αυτό, ότι έχουμε κι εμεί ανησυχίε, ε, ειδικά σε ό,τι αφορά τι αυστηρέ διατάξει για την οδηγία για του οικοτόπου, οπότε θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά μέχρι να λάβουμε την απάντηση από τον Αμένο Βασίλειο και τι αρχέ του. Ε, και φαντάζομαι ότι θα περιμένουμε μετά την Κομισιόν να λάβει απάντηση για το κατά πόσο πληρούνται οι προποθέσει, οι υποχρεώσει ή αν πρέπει να ξεκινήσει, ε, να συνεχιστεί μάλλον η διαδικασία επί παραβάση. Αυτό προτείνω εγώ. Ευχαριστώ και του αναφέροντε για την παρουσίασή του. Είναι πάντα δύσκολο ένα τόσο περίπλοκο και ε, τεράστιο θέμα να το παρουσιάσεις μέσα σε λίγα λεπτά. Χαίρομαι όμως γιατί πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που ακούσαμε. Äh, ναι, Πρόεδρε. Και εγώ θα συμφωνήσω. Αν κατάλαβα καλά, ε, ο σχεδιασμός έχει ε, ανακληθεί. Οπότε δεν θα δημιουργηθεί, δεν θα κατασκευαστεί παρακαμπτήριο. αν κατάλαβα σωστά. Ε, Βέβαια είναι πολύ σημαντικό το θέμα γιατί είναι όντως ευλογημένος αυτός ο τόπος και ε, μιλούμε για πάρα πολλά είδη ε, νυχτερίδων που θα πρέπει να προστατευτούν οπότε θα δούμε κατά πόσο μπορεί να, κατά πόσο εφαρμόζεται σωστά από τις αρχές της Βρετανίας η οδηγία. Όντως δεν έχει νόημα να κλείσουμε την αναφορά οπότε ε, φαντάζομαι ότι και η Κομισιόν το ίδιο, τον ίδιο σκοπό έχει, οπότε γι' αυτό προτείνει να το ερευνήσει περαιτέρω. Συμφωνούμε λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Χαίρομαι που θα το ερευνήσει περαιτέρω η Κομισιόν ε, και θα περιμένουμε τους δύο μήνες για να λάβει η Κομισιόν τις, αποφάσεις, τις απαντήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και να έρθει σε επαφή μαζί μας. Δεν θέλει να παρέμβει κάποιος άλλος. Ωραία. Οπότε παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά όσο θα περιμένουμε και τις απαντήσεις από τις Βρετανικές Αρχές. Πάμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα. Άρθρο, ε, σημείο συγγνώμη 14, ε, αναφορά 632 του 2008 του Robert B. Drone. Ο κύριος Σμίτσεκ είναι εδώ και θα του δώσουμε το λόγο για να παρουσιάσει την αναφορά. Seems, uh, I'm the last one here to, so I Φαίνεται ότι είμαι ο τελευταίος, οπότε θα είμαι και σύντομο. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε τον ε, λόγο, ευχαριστώ που με επιτρέπετε να παρουσιάσω την αναφορά μας. Είναι ε, μεγάλη ημέρα σήμερα, είναι μεγάλη χαρά για την ε, κοινότητά μας να μπορεί να παρουσιάσει την αναφορά εδώ μπροστά στο Κοινοβούλιο. Η αναφορά που ξεκίνησε από τη δική μα οργάνωση από το 2008 θέτει συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία κατά τη δική μας άποψη παραβιάζουν την ευρωπαϊκή ελευθερία κίνησης, καθώς επίσης και τα βασικά δικαιώματα της ιδιωτική ζωής και της οικογενειακής ζωής. Η δική μας αναφορά ε, αφορά περιπτώσεις όπου οι πολιτικές αρχές αρνούνται να δώσουν το, τα πιστοποιητικά για τις άδειες γάμου σε Πολωνούς ε, πολίτες που θέλουν να ε, να κάνουν γάμο με, σε, άλλες, σε άλλα με άτομα του ίδιου φύλου η τα μέλη της, ε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής. Όπως τα γνωρίζετε, η Πολωνία είναι μία από τις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αναγνωρίζει τους, ε, τις σχέσεις ιδίου φύλου και δεν δίνει κανένα δικαίωμα στα άτομα που αποτελούν τη σχέση αυτή, ούτε οικονομικής ούτε οικογενειακής φύσης. Από τότε που η Πολωνία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί από τους ομοφιλόφιλους ε, της ε, ε, Πολωνίας μετακόμισαν, έφυγαν από τη χώρα και ξεκίνησαν ή συνήψαν σχέσεις με αλλοδαπούς. Οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες, νομικά τουλάχιστον, αναγνωρίζουν τις σχέσεις ιδίου φύλου και ζητούν τα δύο αυτά άτομα να αποδείξουν ότι δεν είναι ήδη παντρεμένα που είναι προϋπόθεση για να μπορέσουν να παντρευτούν ή για να μπουν σε μια καταχωρημένη νομική, ε, νομικής φύσεως ε, σχέση. Ε, οι πολιτικοί πολίτες μπορούν να λάβουν αυτά τα έγγραφα από τα Μητρώα της Πολωνίας. Αλλά δυστυχώς οι πολωνικές αρχές αρνούνται να εκδώσουν τέτοια πιστοποιητικά για τους Πολωνούς πολίτες που θέλουν να λάβουν αυτά τα πιστοποιητικά γάμου ώστε να τα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν μία, ένα γάμο ιδίου φίλου σε άλλο κράτος. Γιατί λένε ότι δεν υπάρχει βάση, μια από το πολωνικό νομικό σύστημα δεν αναγνωρίζει και δεν γνωρίζει τέτοιους θεσμούς, όπως αυτός του ε, γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου. Ταυτόχρονα οι Πολωνοί πολίτες που θέλουν να κάνουν γάμο με άτομα του άλλου φίλου μπορούν να πάρουν τέτοια προστοποιητικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Λαμβάνοντα λοιπόν υπόψη αυτή την ε, κατάσταση, θεωρούμε ότι ο μόνος λόγος που γίνεται αυτή η άρνηση είναι η, ε, ο σεξουαλικό προσανατολισμός, ο προσανατολισμός των ετούντων που ζητούν από τις πολωνικέ αρχές να εκδώσουν τέτοια έγγραφα ε, που, χρειάζονται από τις, που τα χρειάζονται οι ξένες οι αρχέ. αρχές. Η κοινότητά μας έχει λάβει πάρα πολλά παράπονα από ομοφιλόφιλους που προσπαθούν να συνάψουν ε, σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τι κάτω χώρε, τη Σουηδία ε, και όλοι δεν, και σε κανένα δεν δόθηκε η άδεια. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά που λαμβάνουμε εμεί, αλλά είναι ε, μεγαλύτερη ευρείας εμβέλεια στο φαινόμενο αυτό. Θεωρούμε ότι ε, υπάρχουν μεγάλα ισχυρά επιχειρήματα για να ε, δοθούν αυτές οι, αυτά τα έγγραφα από τις πολωνικές αρχές για τους, ε, για τους Πολωνούς πολίτες που θέλουν να εξασκήσουν το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και που θέλουν να συνάψουν γάμο ιδίου φίλου σε άλλη χώρα. Υπάρχει και το άρθρο 20 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων πολιτών να κινούνται και να εγκαθίστανται, να εγκαθίστανται ελεύθερα στην ε, στα κράτη-μέλη, στην ε, επικράτεια των κρατών μελών, κατά τη γνώμη μας. Η πρακτική αυτή των, πολιτικών αρχών, των, πολε, των αρχών ε, αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος της, ε, του σεβασμού της οικογενειακής ζωής, που, για το οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εκδώσει και αποφάσεις. Θεωρούμε ότι αυτές οι πρακτικές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Θεωρούμε ότι παρόλο που οι εθνικές αρχές και οι πρακτικές που ακολουθούν σε ό,τι αφορά την έκδοση αυτού του, αυτών των πιστοποιητικών δεν εμπίπτουν στο ε, πεδίο εφαρμογή της ε, Ευρωπαϊκής αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη όταν εξασκούν τι αρμοδιότητές του, μπορούν να παραβλέπουν τις γενικότερε υποχρεώσει που προκύπτουν από τι ευρωπαϊκέ Συνθήκες. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το δικαίωμα για το σεβασμό της οικογενειακής ζωής προστατεύεται από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία ε, εξασφαλίζονται στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ε, υπεγράφηκε στη Ρώμη το 1950 και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, και την ομολογία του προστατεύονται και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θεωρούμε ότι αυτή η πτυχή δεν μπορεί να παραβλέπεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όταν αξιολογούν το πρόβλημα που παρουσιάζεται σήμερα στην αναφορά μας, ειδικά σε ό,τι αφορά την, ε, πρόσβαση, την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Σύμβαση. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ροντρίγκο Μπάλεστερ, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρο μου. Ευχαριστώ και τον αναφέροντα για την αναφορά αυτή που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης. Όντως, ε, καταδικάζουμε την κατάσταση αυτή που περιγράφει ο αναφέρον, όμως νομικά μιλώντας, το θέμα αυτό που είναι θέμα ε, πράξεων ε, πιστοποιητικών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η οδηγία όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία έχει να κάνει με την είσοδο, την κυκλοφορία, αλλά δεν έχει να κάνει με το γάμο ή τις προϋποθέσεις για γάμο. Οπότε αναγκαζόμαστε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν παραβιάζεται η ελευθερία κυκλοφορίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εθνικές αρχές δεν πρέπει να αναγνωρίζουν τους δεσμούς, αλλά όσον αφορά την οδηγία, οι Ευρωπαίοι πολίτες που πάνε σε μια άλλη χώρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την είσοδο σε μια άλλη χώρα. Αναφερθήκατε στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η χάρτα αυτή που είναι νομικά δεσμευτική χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας, εφαρμόζεται όταν πρόκειται για κοινοτική νομοθεσία. Εδώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μπορούμε να επικαλεστούμε τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και μελετάει το θέμα των αστικών δικαιωμάτων για να δει μήπως μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Παρόλο λοιπόν που εξετάζουμε ιδιαίτερη συμπάθεια το θέμα αυτό της αναφοράς, δυστυχώς δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι γι' αυτό. Γιατί δεν είναι θέμα Ευρωπαϊκής Θαγένειας. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν με εκπλήσουν αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εδώ δεν το λέω προσωπικά για εσά, εσεί βέβαια εδώ μεταφέρετε ένα μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα με χίλια ζόρια αναγκαζόταν να κάνει το σωστό. Και όταν πρόκειται για θέματα γάμου, αστικών δικαιωμάτων κτλ. Είναι θέμα κρατών μελών, λέει. Και εδώ Θέλω να ευχαριστήσω τον αναφέροντα βέβαια που ήρθε. Εδώ θα μπορούσε κάτι να κάνει. Όμως, τι πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε αυτό το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης. Αν κάποιο κράτος μέλος πρέπει να δώσει ένα χαρτί που λέει ότι δεν είσαστε σε έναν επίσημο δεσμό μέσα, αν δω εδώ αυτό το χαρτί, είναι ότι σας δυσκολεύει να φτιάξετε ένα τέτοιο δεσμό σε μια άλλη χώρα μέλος. Αν λοιπόν σας αρνούνται αυτό το δικαίωμα, πώς θα μπορέσετε να επωφεληθείτε από τα δικαιώματα που έχετε ως Ευρωπαίος ο πολίτης, εφόσον δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόν τον δεσμό σε μια σχέση ε, καταχωρημένης συμβίωσης ή σε ένα γάμο με άτομο του ίδιου φύλου. Εδώ λοιπόν έχουμε τα επιχειρήματα της νομολογίας που είναι το δικαίωμα σε οικογενειακή ζωή. Αν θέλει κανείς να έχει οικογενειακή ζωή και βέβαια η οικογένεια έχει πολλούς ορισμούς. Εσείς αναφερθήκατε στον κανονισμό του 2004 που αναφέρει οικογένειες Και εδώ περιλαμβάνονται και οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου. Αν λοιπόν, και ας τη βάλουμε στην πάντα αυτή την οδηγία για λίγο, γιατί όσον αφορά αυτήν έχετε δίκιο, έχει να κάνει με την επανένωση μελών μιας οικογένειας. Πάντως το δικαίωμα στην οικογένεια σημαίνει ότι όταν έχετε μια οικογένεια σε ένα κράτος μέλος που αναγνωρίζετε επίσημα, έχετε καθήκοντα και υποχρεώσεις που νόμιμα επιβάλλονται και προσφέρονται. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δύο άνθρωποι έχουν μια σχέση καταχωρημένης συμβίωσης και εγώ σε τέτοια περίπτωση είμαι, σας το λέω δηλαδή. Λοιπόν, αν στην πλατεία του Λουξεμβούργου με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, ή σε κάποια στη ε, πλατεία κτλ ε, άνθρωπος με τον οποίο έχω σχέση μπορεί να πει, έχει δικαίωμα να πει αν ε, εγώ πρέπει να ζήσω σε κόμμα ή να μου σταματήσω το μηχάνημα κτλ. Αν όμως ήμουν πόλονός και μου είχαν αρνηθεί αυτό το χαρτί οικογενειακής κατάστασης, τότε ο φίλος μου δεν θα μπορούσε να παρέμβει, δεν θα είχα δικαίωμα να έχω οικογενειακή ζωή σε εκείνη τη χώρα, οπότε ότι αναφέρει το άρθρο 8 τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα ίσχυε. Υπάρχει και το άρθρο 6 και το άρθρο 7 τη ηθίκη τη Ρώμη που λέει ότι η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι κοινοτική νομοθεσία. Οπότε, ότι δεν σέβεται αυτό το νόμο, τον παραβιάζει. Και με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε και την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που επίσης εφαρμόζεται και ισχύει εδώ και μιλάει για δικαίωμα σε οικογενειακή ζωή. Τέλος, και ξέρετε κύριε Πρόεδρε, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι αστικές ελευθερίες είναι πράγματα που με παθιάζουν, θα μπορούσα να μιλάω για αυτά με τις ώρες. Τέλος, κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι ε, δεδομένης της του Άμστερνταμ που μιλάει για την ευρωπαϊκή κοινότητα, η αρχή της μη διάκρισης περιλαμβάνεται στη συνθήκη όταν πρόκειται για φίλο, ηλικία, ε, γενετήσιους προσανατολισμούς κλπ. που αναφέρονται στο άρθρο 13 της συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 19 και ενισχύεται με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όμως και κάτι άλλο είναι η αρχή της μη διάκρισης βάσει της εθνικότητας. Αν λοιπόν επειδή έχει τη μία την άλλη εθνικότητα, το κράτος μέλος σου, επειδή είσαι πολίτης του, σου αρνείται ένα έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει και μπορεί να σε βοηθήσει να χαρείς των δικαιωμάτων σου, αυτή είναι μια διάκριση βάσει της εθνικότητας. Γιατί είναι η εθνικότητά σου που σε ένα άλλο κράτος μέλος χρησιμοποιείται για να υπονομεύσει ένα δικαίωμά σου. Έχω δει και τη νομική γνωμοδότηση που έχει ετοιμαστεί εκ μέρου των ε, αναφερόντων, θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το διαβάσει. Εγώ θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή, γιατί όπως είπε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και χαίρομαι γι' αυτό, εξετάζει το ρόλο που παίζουν οι αρχές στην περίπτωση τέτοιων πιστοποιητικών και γι' αυτό θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Και βάσει και των συνθηκών στις οποίες αναφέρθηκα, και βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πολλών άλλων που αναφέρονται σε αυτό το άγραφο. Να μείνει ανοιχτή παρακαλώ αυτή η αναφορά. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Κάσμαν ήταν σαρωτικός και όσον αφορά την νομική πλευρά της υπόθεσης και όσον αφορά την ουσία άρα εκ των πραγμάτων μένουν ε, ελάχιστα πράγματα να υποστηρίξει οποιοδήποτε άλλος. Ε, αυτό που σκέφτομαι ακούγοντας την ε, πολύ καλά τεκμηριωμένη αναφορά, ακούγοντας επίσης την πολύ προσεκτικά διατυπωμένη απάντηση της Επιτροπής, είναι ότι εδώ αντιμετωπίζουμε το εξής θέμα. Χρησιμοποιούμε τις οδηγίες, τους νόμους, τις νομοθεσίες αλλά κάρτα. Τις χρησιμοποιούμε δηλαδή κατ' επιλογήν. Όταν μας βολεύει ως Κομισιόν διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής. Όταν δεν μας βολεύει ή δεν θέλουμε να ταράξουμε ισορροπίες, στενεύουμε το πεδίο εφαρμογής και οδηγίας. Αυτό είναι κάτι που δεν μου αρέσει και θα ήθελα πραγματικά να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε κρατώντας ανοιχτές υποθέσεις όπως αυτή για την οποία συζητούμε τώρα. Διότι αισθάνομαι ότι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να παλεύουμε προς όφελος των λαών της Ευρώπης και των πολιτών της Ευρώπης είναι η έκφραση της αλήθειας. Ο άνθρωπος αυτός από την Πολωνία είπε αλήθεια. Ζήτησε πραγματικά αυτό το οποίο ήθελε. Ήθελε να τελέσει ένα γάμο με έναν άνθρωπο ιδίου φίλου. Θα μπορούσε κάλλιστα, εφόσον επιθυμούσε τη σύναψη του γάμου σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης, να μην δηλώσει το φίλο. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα έτσι όπως έχουν, να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια, να δεχόμεθα την αρχή της επιλογής, είναι δικαίωμα ανθρώπινο και υπάρχει και κάτι ακόμη. Το θέμα της παρέμβασης ή μη παρέμβασης. Ένα κράτος μέλος που φέρεται με αυτόν τον τρόπο, εκ των πραγμάτων, έμεσα παρεμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο ασκεί διοίκηση άλλο κράτος μέλος είναι και αυτή μια όψη την οποία θα πρέπει να δούμε, να σκεφτούμε. Και κλείνοντας, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιούμε σαν φερετζέ την νομοθεσία για να καλύπτουμε ζητήματα τα οποία δεν έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε με τα νομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Καταλήγοντας, θα ήθελα και εγώ να ενώσω τη φωνή μου με τους συναδέλφους που λένε ότι η αναφορά αυτή καλό είναι να παραμείνει ανοιχτή όχι μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς αλλά για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η κομισιόν και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα νομικά εργαλεία. Ευχαριστώ. Ε, Der Όντως είναι περίπλοκη η κατάσταση και είμαστε έξι παρα και πρέπει και να κλείσουμε, οπότε θα είμαι σύντομο. Η περίπτωση λοιπόν είναι περίεργη γιατί όντως αυτά τα θέματα από τον και του οικογενειακού δικαίου και αυτά είναι θέματα αρμοδιότητα των κράτων μελών και δεν μπορούν να αλλάξουν. Οπότε και δεν θέλουμε και να αλλάξουμε προς το παρόν τουλάχιστον. Αλλά είναι άλλο θέμα το αν ένας άνθρωπος έχει το δικαίωμα να συνάψει ένα γάμο με άτομο του ίδιου φίλου και αν μπορεί να του αρνείται η αρχή τα πιστοποιητικά που χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν για αυτή την περίπτωση μιλούμε εδώ. Ο κύριο Κάσπαν το είπε πραγματικά σαφέστατα, οπότε θα συμφωνήσω απόλυτα με τη δική του αξιολόγηση. Ήταν ε, ε, πολύ συγκεκριμένο και νομίζω ότι όντω πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά αυτή. Δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει πρόσωπο τη Κομισιόν. Σα ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Δύο λόγια για να επιμείνω και πάλι σε σχέση με την ε, κατανόηση της κατάστασης. Πολωνικά ζευγάρια του ίδιου φίλου, λέει, δεν μπορούν να έρθουν σε οποιαδήποτε είδος σύνδεση σε άλλα κρατέ Παρότι παρά τα όσα μπορεί κανείς να αισθάνεται για αυτή την κατάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κομισιόν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη να ενεργήσει μέσα στις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει. Δυστυχώς λοιπόν εδώ δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Φυσικά και πριν έρθουμε εδώ ε, μελετήσαμε την νομική ε, γνωμοδότηση που για μας δεν είναι νομικά βάσιμη και παρά τα όσα μπορεί να πιστεύουμε από νομική άποψη δεν είναι μέσα στι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ δηλαδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την οδηγία 2048 για να προσφέρουμε κάποια λύση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο Κάσμαν. Σύντομα. Ναι, σύντομα. Μία πρόταση απλώς. Δεδομένου ότι εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι αποτελεσματική και ότι η οδηγία 2004 58 μπορεί να ισχύσει λόγω της άρνησης του, δικαιωμά... του δικαιώματος ε, για ελεύθερη ε, επιλογή της κατοικίας. Εγώ προτείνω να μην ανοιχτή αυτή η αναφορά και να έχουμε μια συνάντηση όσο γίνεται πιο σύντομα με την Επίτροπο Ρέντινγκ που νομίζω ότι είναι η αρμόδια για το θέμα, αν και δεν είμαι βέβαιος. Και είμαι σίγουρος ότι και η Επίτροπος Ρέντινγκ θα θελήσει να το συζητήσουμε αυτό ανοιχτά. Ο κύριος Γιάρα. Να πω απλώς ότι εδώ μιλούμε για δύο πράγματα. Ένα είναι το αν ένα κράτος μέλος ε, μπορεί να αναγνωρίσει τους ε, γάμους του δύο φίλους σε ένα άλλο κράτος μέλος και το άλλο είναι αν ένα κράτος μέλος που αρνείται να δώσει έγγραφα σε ένα κράτο μέλος μπορεί όντω να, να το πράττει αυτό. Ε, βέβαια εντάξει τώρα αν πάω εγώ σε μια αρχή και ζητήσω ένα έγγραφο που χρειάζομαι η, η αρχή δεν έχει δικαίωμα να ρωτήσει τι το θέλει στο χαρτί. Εγώ θέλω ένα χαρτί από την αρχή. Οπότε θα ήθελα πραγματικά να κρατήσουμε χωριστά αυτά τα δύο ερωτήματα και όντω να θα συμφωνήσω ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσει. Ωραία. Πιστεύω πω όλοι συμφωνούν με το να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Και η θέση μάλλον αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι ε, κατά πόσο στα όσα αναφέρονται στην αφορά υπάρχει πραγματικά μία πρακτική διακριτική και άρα παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας και επίσης όπως είπε σωστά ο συνάδελφος Γιάρ, εάν υπάρχει περαιτέρω παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Πρόκειται για έγγραφα του... για το πιστοποιητικό μάλλον οικογενικής κατάστασης και δεν βλέπω πού μπορεί να βασίζεται το ότι πρέπει να δώσουμε αιτιολόγηση γιατί ζητάμε αυτό το έγγραφο. Εγώ θα πρότεινα, γιατί πιστεύω πως είναι σκόπιμο όχι μόνο να μην ανοιχτή η αναφορά, αλλά γιατί με βάση αυτή την αναφορά μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις και η πρόταση που έρχεται στο μυαλό μου είναι να σκεφτούμε και να ζητήσουμε μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που να το ζητήσουμε λοιπόν επισήμως μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. για την οδηγία αυτή. Και όταν θα έχουμε τη γνωμοδότηση θα δούμε αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εγώ νομίζω πως δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε από τις πολωνικές αρχές γιατί το κάνουν αυτό, γιατί η απάντηση είναι ήδη στην αναφορά, γίνεται επί τη βάση τη εθνικής του νομοθεσία, την οποία αυτοί εφαρμόζουν πληρέστατα. Αν υπάρχουν τώρα τιολογήσει ε, έγκυρες για να την συμπεριφορά αυτή από την κυβέρνηση τη Πολωνία θα το ακούσουμε. Αλλά αν όχι, διαφορετικά, αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ζητήσουμε και την γνωμοδότηση της ΛΥΜΠΕ. Αυτά εγκρίνεται και νομίζω πως εξαντλήσαμε και την ημερήσια διαταξή μας για σήμερα και να κλείσουμε να τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ.